Συνάδελφοι, θα ήθελα να καθίσετε σας παρακαλώ για να τιμήσουμε την Επίτροπο, την κυρία Φερέρο Βάλτνερ, η οποία ήρθε ακριβώς την ώρα της. Και επειδή έχει και άλλες υποχρεώσεις, μπορεί να μείνει μαζί μας για μία ώρα και 45 λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν όταν ε, ανοίξουμε τη συζήτηση να αρκεστείτε στο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Και θα έχετε δυνατότητα να παρέμβετε για δύο λεπτά. Δεν υπάρχει λόγος ε, να κάνετε μία εισήγηση θα ήταν σκόπο να αποβάλλετε την ερώτησή σας αποκλειστικά για να μας απαντήσει η Επίτροπος. Θα ήθελα εξ ονόματος της Επιτροπής να εκφράσω την ευχαρίστησή μας και να καλωσορίσω την Επίτροπο σε αυτή τη συνεδρίαση. Βεβαίως γνωριζόμαστε πολύ καλά. Υπάρχουν και πολλοί νέοι βεβαίως στην Επιτροπή και θα ήθελα να την ευχαριστήσω γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα δύο εβδομάδες πριν να συναντηθούμε στο Στρασβούργο. Είχαμε έναν ιδιαίτερα επικοδομητικό διάλογο και με την ευκαιρία εκείνη είχαμε συμφωνήσει ότι θα επικεντρωθούμε την επικείμενη αποστολή όπου θα γινόταν συνάντηση με τους εταίρους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα μας μιλήσει λοιπόν για αυτές τις επαφές και για τις εξελίξεις που ανέκυψαν ως προς το Αφγανιστάν, για παράδειγμα, το Ιράν, το Ιράκ, τη Μέση Ανατολή και επ' αυτού του θέματος ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει ορισμένα περισσότερα πράγματα από αυτά που μας έχει κοινοποιήσει ο τύπος. Και ποιος είναι, και, ποιος είναι ο νέος προσανατολισμός της νέας Αμερικανικής κυβέρνησης σε σχέση με τους επικισμούς του Ισραήλ. Ξέρετε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κατάσταση που έχει αλλάξει άρδιν. Ξέρετε ποια είναι και η νέα στρατηγική της Επιτροπής ως προς τη Λατινική Αμερική. Υπάρχει και η επικείμενη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει τις σκέψεις της. Ε, επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο θα σιωπήσω και θα της δώσω το λόγο ευχαριστώντα της άλλη μια φορά για την παρουσία της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι, με αυτή την ευκαιρία θα προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων στην πρώτη μας ε, επίσημη συνάντηση σε αυτό το νέο κοινοβούλιο. Χαίρομαι για την επικείμενη συνεργασία μας ε, τους επόμενους μήνες. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα και μετά θα σας μιλήσω για την ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής που θα εγκριθεί αύριο. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία ήταν η, η παρουσία και ο λόγος του Μπάρακ Ομπάμα στην ε, Γενική Συνέλευση. Μας μίλησε για τέσσερα θέματα που αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος και που επικράτησαν της ατζέντα, δηλαδή τον αφοπλισμό και μη διάδοση πυρηνικών όπλων, ειρήνη και ασφάλεια, κλιματικές αλλαγές και την παγκόσμια οικονομία. Ως προς τη μη διάδοση, ζήσαμε μια ιστορική στιγμή στη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως προς το ψήφισμα για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Είναι πολύ ενθαρρυντικό όταν βλέπουμε πώς κινήθηκαν οι ΙΠΑ πρόσφατα ιδιαίτερα ως προς τις διμερείς ε, διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, κάτι το οποίο δημιούργησε θετικό κλίμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η διάσκεψη αναθεώρησης της ε, μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, το 2010 δηλαδή, θα δώσει καρποφόρα αποτελέσματα. Δυστυχώς η θετική στάση ε, αμαυρώθηκε διότι το Ιράν μας κοινοποίησε ότι έχει αναπτύξει μία νέα μονάδα πυρηνικών όπλων αμφισβητώντας το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα αυτή η συνάντηση στη Γενέβη είναι κρίσιμη σημασίας για να ορίσουμε την απάντηση της διεθνούς κοινότητας και ελπίζω να έχουμε επικοδομητικές αποφάσεις ως προς την ειρήνη και την ασφάλεια. Δυστυχώς η σύραξη στη Μέση Ανατολή ήταν θέμα που προσέλκυσε την προσοχή αυτή τη βδομάδα, ιδιαίτερα ως προς τον τριμερή διάλογο μεταξύ Ομπάμα, Αμπάς και Νετανιάχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το συζήτησε, καθώς και την ε, ευρύτερη κατάσταση με την Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Κλίντον. Και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το όλο θέμα για να έχουμε μια συνεκτική λύση της σύραξης του αραβικού κόσμου, των Παλαιστινίων δηλαδή, με το Ισραήλ. Όλοι ελπίζαμε να επιτύχουμε περισσότερα, αλλά το γεγονός ότι τα δύο συμβαλόμενα μέρη βρέθηκαν μαζί στην ίδια αίθουσα ήταν ένα επικοδομητικό βήμα. Η Υπουργό Εξωτερικών ε, Κλίντον θεώρησε ότι υπάρχουν δυνατότητες για διαπραγματεύσεις κατά τις επόμενες εβδομάδες και ελπίζω να επιτελεστεί πρόοδος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Όπως ήδη ανέφερε, θα πρέπει όλα τα συμβαλόμενα μέρη να ασχοληθούν με το θέμα των δύο κρατών, της σύστασης δύο κρατών, δηλαδή το Ισραήλ και ένα βιώσιμο κράτος της Παλαιστίνης που να συμβιώνουν ειρηνικά. Επίσης γνωρίζετε ότι είχαμε και το κουαρτέτο της Μέσης ε, Ανατολής, την τετραμερή, την Παρασκευή που τόνισε τη σημασία του τριμερούς ε, διαλόγου που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις και όλοι συμφώνησαν ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να επανακινηθεί η συζήτηση. Προτρέψαμε το Ισραήλ να μην προβεί σε επικισμούς, να επιτρέψει την πραγματική ανάπτυξη, τη φυσική ανάπτυξη και να μην προβεί σε προκλήσεις. Παράλληλα, ζητήσαμε από την Παλαιστινιακή Αρχή να καταβάλει προσπάθειες για το δίκαιο και την τάξη και την καταπολέμηση του εξτρεμισμού. Ξέρετε ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι πολύ δύσκολη και χρειάζεται άμεσα ένα ψήφισμα ιδιαίτερα ε, έτσι ώστε να, μπορούν, να μπορεί να υπάρξει ελεύθερη διακίνηση από τα σημεία ελέγχου για ανθρωπιστική βοήθεια, για τρόφιμα και για ιατρικά είδη. Και ελπίζουμε να επανακινηθεί η διαπραγμάτευση. Όλοι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε τα συμβαλώμενα μέρη να βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να παραμείνουν εκεί. Το Πακιστάν ήταν ένα άλλο θέμα συζήτησης, με το Αφγανιστάν, αλλά είχαμε μια ειδική συνάντηση μέσα στα πλαίσια της διάσκεψης κορυφής με το Πακιστάν, τους φίλους του Πακιστάν, έτσι ώστε να τονίσουμε το ότι το Πακιστάν προσπαθεί να προβεί στη σταθεροποίηση της χώρας και την καταπολέμηση του εξτρεμισμού. Το Πακιστάν βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή καταπολέμηση της τρομοκρατίας και βεβαίως αυτό αφορά και τις άμεσα και τις γειτονικές χώρες. Άρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνής κοινότητα τονίσαμε την ε, δέσμευσή μας έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να υπάρχει μία μακροχρόνια λύση καταπολέμησης του εξτραμισμού. Ως προς τις κλιματικές αλλαγές, ο Γενικός Γραμματέας ε, του, των Ηνωμένων Εθνών και με βάση την απόφαση των G20 στο Πίτσμπεργκ θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να επέλθει συμφωνία στην ε, Κοπενχάγη και η δέσμευση της Ιαπωνίας ήταν ύψης της σημασίας διότι συνεισφέρει έτσι ώστε να φτάσουμε σε, σε έναν σε μια απόφαση με διτό στόχο. Όμως πρέπει να επιτελεστεί πολύ μεγάλη ε, προσπάθεια έτσι ώστε οι βιομηχανικές χώρες έτσι ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή ε, μετριασμού, έτσι ώστε να φτάσουμε μεταξύ 2 και 15 ε, δις μέχρι το 2020. Αν υποθέσουμε ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία στην Κοπενχάγη. Ως προς μια βιώσιμη και εξισορροπημένη παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της Κοπενχάγης και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να πείσει και τους άλλους να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο δέσμευσης ως προς την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία μας απασχόλησε και στο Πίτσμπεργκ. Μιλάμε για ένα θέμα ε, που αφορά την, ε, το χρηματοπιστωτικό και τη ρυθμισή του. Πρόκειται για έναν διτό στόχο έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε και τα αίτια της κρίσης, αλλά χρειάζεται συντονισμένη δράση μέσα στα πλαίσια και των στόχων της ε, χιλιετίας. Οι G20 ανέλευαν δεσμεύσεις και στα δύο μέτωπα, αλλά βεβαίως το βασικότερο είναι η εφαρμογή. Και εδώ σε Ευρωπαϊκή Ένωση διανοίγουμε το δρόμο ε, ε, με βάση τις δικές μας πρόσφατες προτάσεις και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πλήρωση αυτών των στόχων. Πέρα από αυτά τα θέματα, Είχαμε και ορισμένα θέματα πυρήνες, όπως ξέρετε μιλήσαμε για την μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα πρέπει να βρούμε μια καινοτόμο λύση. Παράλληλα όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλους τομείς. Επ' αυτού ε, θα πρέπει να πω ότι το θέμα της ισότητας των δύο φύλων επικράτησε τις συζητήσεις και μιλήσαμε για έναν ειδικό φορέα μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Και χρειάζεται η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών. Στην αρχή είχαμε ένα πρόγευμα με την, ε, το ψήφισμα 2025. Στη συνέχεια έχουμε ένα γεύμα υπό την αιγίδα της κυρίας Κλίντον και στη συνέχεια είχαμε μια συζήτηση για τις ε, κλιματικές αλλαγές υπό την ε, αιγίδα του Προέδρου της Λιβερίας. Ως προς το πρόγευμα προωθήσαμε τις, ε, τα δύο ψηφίσματα 1325 και 1820 έτσι ώστε να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων και να προωθήσουμε το όλο θέμα πριν από την ε, μεταρρύθμιση που θα γίνει του χρόνου. Ως προς τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής αύριο το πρωί θα προβώ σε μία ανακοίνωση για τα 10 χρόνια στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Εάν λάβουμε υπόψη το γενικό παγκόσμιο υπόβαθρο και το, την νεαρινή σύνοδο της Μαδρίτης του χρόνου θα πρέπει να σκιαγραφίσουμε τους στόχους, τους απότερους στόχους για μια στρατηγική προς την περιφέρεια αυτή στα επερχόμενα χρόνια. Τη στιγμή που οι διεθνείς συμμαχίες έχουν μεγάλη σημασία για να αντιμετωπίσουμε τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις, θα πρέπει να ενισχύσουμε και αυτή τη συνεργασία με την περιφέρεια. Θα πρέπει λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προσδώσουμε μεγάλη σημασία συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική, να αντιμετωπίσουμε την χρηματοοικονομική ε, κρίση, τις κλιματικές αλλαγές, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας και ελπίζουμε να δοθεί μια νέα όθηση στις σχέσεις μας αποστέλλοντας ένα σημαντικό μήνυμα στους εταίρους, ενισχύοντας τους δεσμούς με τη Λατινική Αμερική και προετοιμάζοντας και την ε, Ισπανική Προεδρία το επόμενο εξαμήνου. κατά πόσο όλα αυτά, δηλαδή η συγκυρία, βοήθησε στην κοινωνική και πολιτική αναβάθμιση της Υπήρου αυτής και θα ήταν σκόπιμο να ορίσουμε, να προβούμε σε μία ανάλυση για τα σχέδια, σχέδια διαπραγμάτευσης ε, σύνδεσης ή εταιρικής σχέσης μάλλον. Νομίζω ότι θα έπρεπε ως Κοινοβούλιο να χαρούμε διότι το χρηματοοικονομικό μέσον που θα έπρεπε να λέγεται μέσο Φερέρα Βάλτνερ βοήθησε ιδιαίτερα την Ήπειρο αυτή. Είναι πολύ φιλόδοξη πρόταση και τέλος θα ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση στην Ονδούρα. Κύριε Επίτροπε, Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Άριας της Κώστα Ρίκα προσπαθεί να διαμεσολαβήσει για μια ειρηνική επίλυση, αλλά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει έτσι ώστε να εξευρεθεί μια δημοκρατική, συνταγματική και ειρηνική λύση για την κατάσταση στην Ονδούρα. Στο δύο λεπτά ακριβώς, μπράβο. Κυρία Μουνίφ, επίσης δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πω ότι βλέπω ο κύριος Σαλαφράνκα γνώριζε για την ανακοίνωση της Επιτροπής, ε, εγώ δεν μπόρεσα να έχω πρόσβαση σε αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, όπως ξέρετε, δύο σε δύο εβδομάδες θα γίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Χίλη και θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και πώς αντιμετωπίσουμε τα βασικά ζητήματα αυτής της διάσκεψης, ιδιαίτερα ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και την βιομηχανική ιδιοκτησία ως προς την κατάσταση στη Χιλή για, και για την ε, γεωργική ανάπτυξη την τεχνολογία και την ε, καινοτομία. Η Χιλή μάθαμε ότι θα ήθελε να ακολουθήσει το Ιαπωνικό ψηφιακό τηλεοπτικό σύστημα μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν ελήφθησαν υπόψη από τη Χιλή. Και μέλος αυτής της Επιτροπής ε, μας ε, μίλησε χτες ο, ο κύριος Μιγκαρέλη, ο Γενικός Διευθυντής Ρέλεξ, για μία συμφωνία πλαίσιο με τη Λιβύη, οποία καλύπτει πολλές πτυχές μέσα στα πλαίσια των διμερών. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι στην ουσία μιλάμε για μία συμφωνία σύνδεση, δυνάμει του άρθρου 133 της Σύνθηκης. Δεν, μου επιβεβαιώθηκε, μας επιβεβαιώθηκε ποια είναι η νομική ε, βάση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μας πείτε εσείς ποια είναι η νομική βάση, έτσι ώστε να γίνεται διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο πιο συχνά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάποιες λεπτομέρειες όπως το τηλεοπτικό σύστημα είναι πιο τεχνικής φύσεως και όχι πολιτικής φύσεως και επομένως δεν είναι το κατάλληλο βήμα εδώ για να θέσουμε αυτές τις ερωτήσεις στην Επίτροπο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Το Κοινοβούλιο έχει στείλει ψήφισμα στο Συμβούλιο σχετικά με το τι περιμένει από τη γενική αυτή συνέλευση. Αναφέρεται εκεί κάτι και για, ε, ε, ε, τη μεταρρύθμιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Περιέχει προτάσεις σχετικά με τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη. Θέλουμε αναθεώρηση του τρόπου εργασίας του συμβολείου Ασφαλείας. Στο Συμβούλιο υπάρχει σημαντική διαφωνία για το θέμα αυτό. Θα σας παρακαλούσα να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση, τι γίνεται στο Συμβούλιο, πόσο, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα, πόσο ικανοποιημένοι ή όχι είσαστε ε, την κατάσταση. Δεύτερον, μας μιλήσατε για το Gender Equality Architecture Reform, την ε, ε, μεταρρύθμιση αυτή όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Υπάρχει η UNIFAM, υπάρχει η UNFPA, υπάρχουν τα προγράμματα για τις γυναίκες του UNDP. Το gender mainstreaming είναι, mainstreaming είναι ένα οριζόντιο θέμα. Δεν φοβάστε ότι με ένα νέο οργανισμό θα έχουμε με δομική ενίσχυση, αλλά ε, επί της ουσίας θα έχουμε αποδυνάμωση στο θέμα αυτό. Και τελευταία παρατήρηση, και θα ήθελα να συμφωνήσω με τη συνάδελφο από τους Σοσιαλδημοκράτε όσον αφορά την ε, Λιβύη. Λιβύη. Ε, χθες ε, ακούσαμε από τον κύριο Μιγκαρέλη σχετικά. Ε, τι μπορείτε να μας πείτε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. δύο λεπτά. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Αναφέρατε ότι αύριο θα παρουσιάσετε μία έκθεση σχετικά με την Λατινική Αμερική. Θα ήθελα ε, να ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι στο Μεξικό είναι δραματική η κατάσταση. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο πριν ε, δύο-τρία χρόνια είχαμε μία ε, έκθεση σχετικά με τις γυναίκες ε, και το θέμα της ατιμορρησίας στο Μεξικό. Θα ήθελα να ακούσω από εσά τι κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση και όσον αφορά τις γυναίκες και τους φόνους που πραγματοποιούνται στο Μεξικό. Επίσης, όσον αφορά τη συνεργασία στον ε, τομέα της ε, προστασίας αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί απειλούνται από την αστυνομία, από συμμορίες κλπ. Και κάτι ακόμα. Υπάρχουν πολλά κράτη της Λατινικής Αμερικής που δεν ε, τηρούν τις ε, συμβάσεις ε, σχετικά με την, τα δικαιώματα των εργαζομένων κλπ. Αυτό συχνά παρουσιάζει προβλήματα στις σχέσεις Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Τι κάνετε για το θέμα αυτό. Και κάτι ακόμα. Διαπραγματεύσεις ε, για τις ε, συμβάσεις ε, ελεύθερου εμπορίου, ιδιαίτερα με τις Ονδούρες. Τι γίνεται εδώ, συνεχίζονται οι προσπάθειες. Ο κανονικός πρόεδρος βρίσκεται στο στην πρεσβεία της Βραζιλίας. Νομίζω ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. 11 δευτερόλεπτα θα μιλήσετε παραπάνω. Ο επόμενος ομιλητής Έτιτς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τρεις γρήγορες ερωτήσεις, λέει ο κύριος Άτκινς. Για το Ιράν, καταρχάς. Τι προσπάθειες καταβάλλονται από τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεργαστούμε με την Κίνα και τη Ρωσία για να τους πείσουμε για την προφανή ανάγκη και αποτελεσματικότητα των κυρώσεων στο Ιράν αν δεν κάνουν αυτό που τους ζητούμε σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Δεύτερον, Υπάρχει γενική αποδοχή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του Αφγανιστάν. Και αν ναι, σημαίνει ότι οι έρευνες από την ομάδα μας αγνοούνται. Και αν έχουν γίνει αποδεκτές οι εκλογές, τι προσπάθειες θα γίνουν για να βοηθήσουμε το Πακιστάν, που όπως είπατε και εσείς επίτροπε, είναι το κλειδί στην όλη διαδικασία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το Πακιστάν. Ε, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουν, ίσως ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τελευταίο σχόλιο για τη Μέση Ανατολή. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν στοιχεία κάποιες παραγωγικής δραστηριότητας <laughs> από πλευράς του Τόνι Μπλερ. Ευχαριστώ τον κύριο Άτκινς. Μας χαρίσατε και κάποια δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Μπενίτα για την εισήγησή σου και η δική μας ομάδα παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών και το πιο προεξάρχον σημείο ήταν η δήλωση του Προέδρου Ομπάμα. Κάτι το οποίο σήμανε μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την προγενέστερη πολιτική των ΗΠΑ. Άρα θα πρέπει να βασιζόμαστε σε πολυμερείς ε, σχέσεις και όχι σε διμερείς. Η κυβέρνηση Bush άφησε έναν πιο ανασφαλή και πιο άδικο κόσμο, διότι δεν τήρησε το διεθνές δίκαιο. Ελπίζω αυτή η ιδέα να προωθηθεί έτσι ώστε να βάλουμε μία τάξη το, η επόμενη σύραξη αφορά την Μέση Ανατολή. Δηλαδή μετά την συμφωνία της ε, Αναπόλεως βλέπουμε ότι η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ δεν τηρεί τους όρους τους οποίους συμφώνησε η προγενέστερη κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι που οδηγεί σε αδυναμία σύστασης Παλαιστινιακού κράτους όπως όριζε η διάσκεψη και η συμφωνία της αναπόλεως. Ως προς την κατάσταση στην Ονδούρα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκαναν το καθήκον τους. Γίναμε ε, ε, αρρωγή και κοινωνή της κατάστασης ε, που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία δήλωση που να καταδικάζει το πραξικόπημα στην Ονδούρα. Ελπίζω να επανορθώσουμε την κατάσταση. Ο Μιτσελέτη, ο πραξικοπηματίας, σε 10, σε μέρες θα πρέπει να ορίσει πώς έχει η κατάσταση σε σχέση με την πρεσβεία της Βραζιλίας, όπου έχει κλειστεί ο νυν πρόεδρος. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε τι θα γίνει με την ε, πρεσβεία της Βραζιλίας, έτσι ώστε να δράσουμε τάχιστα. Την επόμενη εβδομάδα ο Ερνέστο Ρέγες θα είναι εδώ που είναι μέλος της ε, αντίστασης, της πολιτικής αντίστασης, αστικής αντίστασης στη χώρα και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η στάση σας. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε εκτός χρόνου. Πέτερινγκ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συμμερίζεστε τη θέση ότι αν δεν υπάρχει ειρήνη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, αυτό θα έχει σοβαρές ε, συνέπειες ε, στη σχέση μας με τον αραβικό κόσμο και στην επιτυχία του διαλόγου των πολιτισμών. Αυτή είναι η ερώτησή μου Έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Ε, μάλλον θέλουμε ε, δύο ανεξάρτητα κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνη, ε, ως προϋπόθεση για τη σχέση μας με τον αραβικό κόσμο. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε τι κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη για την ε, διαδικασία ειρήνης ε, στη Μέση Ανατολή. Ο συνάδελφος Σαλαφράγκα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Αναφέρατε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών ε, τι θα μπορούσε να περιέχει ένα τέτοιο ψήφισμα. Όταν κάποιος έχει αναλάβει νομικές υποχρεώσεις και δεν τις στηρεί, ε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Bene, allora, finito il primo round. Πολύ ωραία. Τελείωσε ο πρώτος γύρος ε, ερωτήσεων και θα δώσουμε το λόγο τώρα στην Επίτροπο. Φέρερο Βάρτινερ για να μας απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με κάποιες και θα συνεχίσω. Καταρχάς, η πρώτη ερώτηση του κ. Σαλαφράγκα για το Ιράν. Στους διάφορους γύρους που είχαμε, καταρχάς μία στο G8 και έναν άλλο γύρο στο G20, το θέμα του Ιράν προφανώς τέθηκε και ήταν ψηλά στην ατζέντα μας. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε σε αυτή τη φάση. Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι έχουμε μια διτή προσέγγιση. Ξέρετε ότι ο Χαβιέρ Σολάνα θα πάει 1η Οκτωβρίου στη Γενέβη. Έχει μια σειρά από συνεδριάσεις και ξέρετε ότι η νέα Αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι αν οι Ιρανοί ε, πάρουν την, την ανοιχτή παλάμη, όπως είπε και ο Ομπάμα, τη δεχτούν, τότε υπάρχει δυνατότητα διαλόγου. Υπάρχει περίπτωση διαλόγου, αλλά τώρα απόκειται στους Ιρανούς να δεχτούν το διάλογο. Όπως είπα και στην ε, πρώτη παρέμβασή μου, τώρα έχουν επίσημα αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα δεύτερο ε, εργοστάσιο για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Μυστικό εργοστάσιο. Η κατάσταση είναι δύσκολη, προφανώς. Επομένως, τη στιγμή που εμείς διενεργούμε το διάλογό μας, θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε το ενδεχόμενο ενδυνάμωση των κυρώσεων. Και ο πρόεδρος Μετιέντεφ της Ρωσίας ξεκαθάρισε ότι ακόμη και η Ρωσία ήθελε να εφαρμόσουμε μια πιο στεναρή στάση. Μόλις ξεκινήσαμε το διάλογο βέβαια, ίσως είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι αλήθεια ότι η υπομονή κάποια στιγμή θα εξατληθεί για το διάλογο. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση για το θέμα του Ιράν. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τη Λατινική Αμερική. Έχουμε 10 χρόνια εταιρικής σχέσης. Χαίρομαι που τα έζησα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι δεν μπορώ να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες αυτής της ανακοίνωσης. Δεν λειτουργούμε έτσι. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε καταρχήν την ε, ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα θα μας δώσει την ευκαιρία να δουλέψουμε με πιο ενδελεχή τρόπο με τη Λατινική Αμερική. Θέλουμε καλύτερο πολιτικό διάλογο και για τομεακά θέματα. Ξέρετε όλες τις μοντέρνες προκλήσεις που υπάρχουν, το, την ασφάλεια της ενέργειας, το, την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα θέματα προφανώς Επίσης, είπατε ότι θα δημιουργηθεί ένα ειδικό, κάποια ειδικά θεμέλια, ελπίζουμε τουλάχιστον να δημιουργηθούν στην ε, Σύνοδο Κορυφής της ε, Μαδρίτης, και θα υπάρξει και ένα συγκεκριμένο μέσο ε, για τη χρηματοδότηση για όλα αυτά τα θέματα, ενεργειακή ασφάλεια, ε, κλιματική αλλαγή. Σας παρακαλώ όμως καταλάβετε ότι δεν μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες, γιατί αλλιώς ε, δεν πρόκειται να έρθει κανένα δημοσιογράφος όταν ανακοινώσω την ανακοίνωσή μου. Θα σας τα έχω πει όλα για την Ονδούρα. Κάποια παρατήρηση γίνεται εκτό μικροφώνου. Ευτυχώ ή δυστυχώς υπάρχουν δημοσιογράφοι. Ε, και εδώ, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Αν συνεδριάζαμε και κλεισμένο το θηρό θα σα έλεγα περισσότερα, αλλά δυστυχώς είναι εδώ οι δημοσιογράφοι για την Ονδούρα. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι οτιδήποτε έχει συμβεί, οτιδήποτε και αν έχει συμβεί, η μόνη πραγματική λύση είναι ο διάλογος σαν Χωσέ και η πρόταση του Όσκαρ Αρίας. Ίσως προκύψουν εκλογές. Αλλά αν έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα από αυτό το διάλογο, θα μπορούσαμε να δεχτούμε τις εκλογές. Ξέρω βέβαια ότι με τη νέα κατάσταση τώρα, όπου ο πρόεδρος Σελάια έχει καταφύγει στην ε, πρεσβεία της ε, Βραζιλίας, τα πράγματα έχουν περιπλακεί περαιτέρω. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά είμαστε αλληλέγγυοι, με όσους θέλαν να διώξουν τους ε, πρέσβεις. Ή μάλλον να τους ε, στείλουν πίσω. Αλλά τώρα δεν μπορούν να τους στείλουν πίσω. Πάντως, ε, σε αυτή την ειδική συνάντηση ε, είπαμε ότι θα πρέπει να δουλέψει ο διάλογος σαν Χωσέ και να βρούμε κάποια λύση. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές κάποια benchmarks. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τη Χιλή τώρα. Η Χιλή είναι μία από τις χώρες ε, όπου οι σχέσεις μας πλαταίνουν και βαθαίνουν. Ε, υπάρχει πρόοδος. Και δουλεύουμε, δουλεύουμε στα πλαίσια μιας συνεργασίας για την ανάπτυξη η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτή η συμφωνία εστιάζει κυρίως στην ενέργεια και κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στην εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε ότι οι στενές μας σχέσεις είναι πραγματικότητα και ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά με τη Χιλή. Γιατί η Χιλή μας προσεγγίζει όλο και περισσότερο. Και εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο, όσο μπορούμε. Την παραμονή της συμφωνίας μεταξύ της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα βρεθεί κάποια λύση. Για τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά πρότυπα. Δυστυχώς αυτό το παιχνίδι το χάσαμε. Το κέρδισε η Βραζιλία. Εγώ δούλεψα πάρα πολύ με διάφορες χώρες, με τους υπουργούς εξωτερικών και με τους αρμόδιους υπουργούς. Αλλά ξέρετε, ότι το πρότυπο στη Βραζιλία είναι η Τζαμπάν, η, Ιαπωνία. Και η Ιαπωνία έκανε πολύ ισχυρό ε, λόμπι σε όλη την περιοχή και τελικά οι Χιλιανοί αποφάσισαν ότι προτιμούν την περιφερειακή λύση. Αλλά βέβαια αυτό δεν ήταν η καλύτερη λύση για μας. Για τη Λιβύη. Η Λιβύη είναι η μόνη χώρα όπου δεν είχαμε καμία συμβατική συμφωνία και προσπαθήσαμε, και ξέρετε ότι εγώ το υποσχέθηκα, όταν ο Παλαιστίνιος γιατρός και οι Βουλγάρες νοσοκόμες απελευθερώθηκαν, ότι θα το υποβάλω στο Συμβούλιο να πάρουμε εντολή και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό έγινε. Και τώρα ε, το πλαίσιο, η συμφωνία πλαίσιο με τη Λιβύη είναι ένας τρόπος για να ξεκινήσουμε ένα πιο ουσιαστικό πολιτικό διάλογο και συνεργασία για τα οικονομικά, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και για τα θέματα της Αφρικής. Ξέρετε πολύ καλά τα θέματα ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικά και είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε, ε, να συμφωνήσουν οι Λίβοι κυρίως ε, σε μια συμφωνία επανιστοχής. προκειμένου να υπάρχει κάποια, κάποιο τροχοπέδι στο θέμα των προσφύγων. Για την νομική βάση τώρα είναι πολύ πρόωρο να προσδιορίσουμε την νομική βάση της μελλοντική συμφωνίας. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων και ανάλογα με το περιεχόμενο της συμφωνίας θα κάνουμε μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο. Και σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον επικυρωθεί και η Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο ρόλο να παίξει. Προς το παρόν ε, αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι θέμα προσφύγων και θέμα ε, συμφωνίας επανεισδοχής. Αυτό μας δυσκολεύει τα πράγματα. Κατά λοιπά όμως, οι διαπραγματεύσεις δουλεύουν αρκετά καλά. Για την ε, μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλα όσα είπατε κύριε Λάμστορφ, αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα θέλαμε να βρεθεί λύση. Ξέρουμε βέβαια ότι στο Συμβούλιο, και σας λέω τη γνώμη μου μια και με ρωτάτε, δεν υπάρχει κοινή θέση. Νομίζω ότι οι θέσεις των κρατών μελών δεν έχουν εξελιχθεί. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη δέχονται τώρα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη εκπροσώπηση το είδαμε ήδη στο, στο G20 ότι υπάρχουν τα ψήγματα κάτι, μια τέτοια ιδέα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Και είναι κρίμα, γιατί πολλές από αυτές τις χώρες θεωρούν ότι είναι αποκλεισμένε. Και επομένως μερικές φορές δεν είναι τόσο πρόθυμες όσο θα έπρεπε. Για το άλλο θέμα που θέσατε για τις γυναίκες. Εγώ συνεργάστηκα πολύ με αυτούς τους φορείς, με την κυρία Μεγκύρο, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, της UNIFAM κτλ. Νομίζω ότι εξαρτάται από την προσωπικότητα που θα ηγηθεί αυτής της δομής. Γιατί αυτό που θέλουμε, θέλουμε ο 18-20 και ο 13-25 να εφαρμοστούν. Υπάρχουν τα ψηφίσματα, είναι καλά, όλοι είμαστε υπέρ, τώρα θέλουμε να υλοποιηθούν. Για το θέμα των λύσεων μετά τις σειράξεις, Φερρυπίν, ή για τα θέματα των διαπραγματεύσεων. Πού είναι οι γυναίκες διαπραγματευτές, σχεδόν υπάρχουν. Στην Αφρική, ας πούμε στη Ρουάντα, πάνω από το 50% της κυβέρνησης, ακόμη και του Κοινοβουλίου, νομίζω είναι γυναίκες. Μετά τις συγκρούσεις, Κατάλαβαν αυτοί οι λαοί ότι πρέπει να δώσουν δύναμη και εξουσία στις γυναίκες. Βοηθάμε τις γυναίκες να δημιουργήσουν το απαραίτητο δυναμικό. Ξέρω ότι κάποια τα κράτη-μέλη, όπως το δικό μου, ας πούμε, το έκαναν. Εγώ ως υπουργό Εξωτερικών είχα βοηθήσει πολύ και χαίρομαι να βλέπω γυναίκες στις επάλξεις. Γυναίκες με εξουσία. Επομένως, δεν είμαι κατά αυτή τη δομή στο βαθμό που συντονίζει όλες οι υπόλοιπε. Και αυτό είναι σημαντικό για, τον, για την ομιλία του Καντάφη. Τι να σας απαντήσω, δηλαδή θέλετε. Κυρία Λούνατσεκ, για το Μεξικό. Είχαμε έναν μακρύ διάλογο με το Μεξικό και για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε μιλήσει για τους φόνους γυναικών, για την ατιμορρησία και το Μεξικό πράγματι έχει κάνει πολλά. Έχουμε συνεργαστεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τους έχουμε βοηθήσει ε, για βελτίωση της αστυνόμευσης. Συνοδεύουμε λοιπόν την όλη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς όμως Υπάρχει ακόμα ατιμορρησία σε μεγάλο βαθμό. Ακούμε συνέχεια από τους Μεξικανούς ότι αυτό συμβαίνει κυρίως στις συνοριακές περιοχές. Όπως ξέρετε υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. Το Μεξικό συνεχίζει τον αγώνα κατά του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε και μάλιστα ε, ε, διαθέτουμε περισσότερους πόρους για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού. Το ίδιο ισχύει για το ILO, το Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Δεν γίνονται σεβαστοί σεβαστεί οι κανόνες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε όλες τις χώρες. Ε, πρέπει όμως να συνεχίσουμε σταθερά το διάλογο αυτό και συχνά όπως ε, στην Κεντρική Αμερική, και αυτό ήταν ένα από τα θέματα κλειδιά, πρέπει να μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι τελικά έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα, όχι όμως όλα όσα θέλαμε. Όσον αφορά την Κεντρική Αμερική και την Ονδούρα, ξέρετε ότι θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεών μας με την Κεντρική Αμερική. Το θέμα υπάρχει. Μόλις λυθεί το θέμα με τις μπανάνες και ελπίζω στην Γενέβη οι συζητήσεις που έχει αυτή τη στιγμή ο Επίτροπος Εμπορίου μας να ε, καταλήξουν θετικά. Τότε θα επανέλθει το θέμα της Ονδούρας και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, διάφορες λύσεις το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει. Μπορεί να αποκλειστεί η Ονδούρα ή να υπάρξει κάποια ρεαλιστική θέση. Για παράδειγμα, να συμμετέχει σε τεχνικό επίπεδο κάποιος, ε, ένα πρώην μέλος που να ε, γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση. Ως προς το Ιράν νομίζω ότι ήδη απάντησα. Ήταν η ίδια ερώτηση που ακούσαμε και πριν. Πιστεύω ότι έχουν γίνει προσπάθειες, κύριε Άτκινς, ώστε και η Ρωσία και η Κίνα να συμμετέχουν. Τώρα όμως είναι χρόνος για διάλογο και θα πρέπει να δούμε μετά αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Ως προς το Αφγανιστάν και το Πακιστάν δεν έχουν γίνει ακόμα απόλυτα αποδεχτέ οι εκλογές. Σημαντικό είναι ότι καταρχήν είχαμε αποστολή παρατηρητών ε, στις εκλογές. Έπρεπε να το ε, αναλάβω αυτό ε, σε πολύ δύσκολη εποχή. Ο πρώην συνάδελφός σας, στρατηγό Μοριών, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήμουν ιδιαίτερα περήφανη γι' αυτόν. Από την άλλη όμως μας εξαπάτησαν. Ζήτησα λοιπόν από τους Αφγανούς να τηρήσουν τουλάχιστον τους δικούς τους κανόνες, τους δικούς τους νόμους. Δηλαδή, να έχουν Επιτροπή Παραπώνων για τις εκλογές και την Επιτροπή Εκλογών. Και τώρα θα πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει κάθε προσφυγή που κατεγράφει. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Μετά όμως θα πρέπει να λάβουμε απόφαση αν δεχόμαστε το αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής αυτής. Και κατόπιν θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την αφγανική κυβέρνηση, διότι αυτό είναι το επόμενο σημαντικό ερώτημα. Ε, η στρατηγική μας, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τη στρατηγική αυτή. Θα ξέρετε ότι υπάρχει καινούριο έγγραφο της ε, Κομισιόν ε, και του Συμβουλίου για το Αφγανιστάν που έχει να κάνει με την ανάπτυξη κανόνων την ε, μείωση της ε, παραγωγής ε, ναρκωτικών, την οικοδόμηση δυναμικού, την δημιουργία του κράτους κλπ. Και ως προς το Πακιστάν. Να πω για το Πακιστάν, πολύ σωστά είπατε και εγώ το ανέφερα, ότι το Πακιστάν είναι μία από τις χώρες κλειδιά. Επίσης ε, έχουμε παρακολουθήσει εκεί τις εκλογές. Ε, ο κύριος Κάλερ ήταν εκεί ε, παρατηρητής μας σε δύσκολες συνθήκες. Έχουμε, λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση που να κάνει ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι Υπήρχαν επιτυχίες ε, ως προς τις αναταραχές ε, στις ε, περιοχές των Ταλιμπάν, τώρα όμως θα πρέπει να παράσουμε κάθε δυνατή υποστήριξη για να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Η Κομισιόν έκανε, κατέβαλε κάθε προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό σε όλους τους τομείς όπου είναι απαραίτητο. Εκπαίδευση, οικοδόμηση δυναμικού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις χώρες αυτές, δημιουργία του κράτους, ε, βοήθεια στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας, σε ανάπτυξη κανόνων κλπ. Ως Επίτροπος για τις εξωτερικές σχέσεις, Βλέπετε ότι συχνά αυτό που μου λείπει είναι η χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα χρήματα για να κάνουμε όλα αυτά τα θέματα που είναι τόσο σημαντικά για όλους μας. Το λέω αυτό διότι στο μέλλον θα πρέπει να ε, σκεφτούμε το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι νωρί ακόμα, αλλά ε, είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου όταν μιλάμε για τα θέματα αυτά. για τη Μέση Ανατολή. Αναφέρατε συγκεκριμένα τον Τόνι Μπλερ. Να πω ότι υποστηρίζω την, ε, τον Τόνι Μπλερ διότι πιστεύω ότι το οικονομικό κομμάτι της δουλειάς του, και αυτή είναι η εντολή του άλλωστε, είναι πολύ σημαντικό. Και γνωρίζετε τι απαιτείτε. Το ξέρω διότι είμαι σε συνεχή επαφή μαζί του. Οι συνεργάτες μας όμως κάνουν, κάνουν το ίδιο πράγμα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε προγράμματα. Θέλουμε να εξαλείψουμε τα εμπόδια. Είναι δύσκολη δουλειά, πολύπλοκη. Κάποια πράγματα όμως έχουν λειτουργήσει. Στη Δυτική Όχθη έχουμε ανάπτυξη 7%, πράγμα που δείχνει στου Παλαιστινίου ότι υπάρχει ελπίδα μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης ε, αν ε, ασχοληθούν με τα θέματα ασφάλειας. Και αυτό μπορεί έτσι να ενισχύσει τον ε, πρόεδρο Αμπάς. Συμφωνώ. Ε, κύριε Πέτερινγκ, στα γερμανικά να πω, έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Αν δεν υπάρχει η ειρήνη, θα έχουμε σοβαρές συνέπειες στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στον αραβικό πολιτισμό και εμάς, αλλά και ε, στο σύνολο της Μέσης Ανατολής σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν είναι υψή τη σημασίας να συνεχίσουμε, και το κάνουμε εδώ και 15 χρόνια, να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε τουλάχιστον να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές. Είναι πολύ δύσκολο, η ε, πολιτική ε, επίκηση συνεχίζεται, δεν υπάρχει συμφωνία για πάυση της πολιτικής αυτής. Ε, συνεχίζονται όμως και οι και οι αμερικανικές προσπάθειες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρούμε μία λύση που θα φέρει τα δύο μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. ελπίζω ότι στις 15 ε, Οκτωβρίου, ελπίζω η 15 Οκτωβρίου να είναι σημαντική ημερομηνία. Εμείς ως ε, κουαρτέτο έχουμε προσανατολιστεί σε αυτή την προσέγγιση και τα ψηφίσματα που αναφέραμε είναι τα ψηφίσματα που αναφέρθηκαν στη δήλωση του κουαρτέτου. Δεν είναι... Ε, ε, είναι μια σειρά ψηφισμάτων, το 242 και άλλα, ε, στα οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία. Θα πρέπει όμως να εποφεληθούμε από την ορμή που έχει δώσει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση και το λέμε αυτό στους Ισραηλινούς αλλά και στον Πρόεδρο Αμπάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ήσασταν πολύ ακριβείς και λακωνικοί ταυτόχρονα. Για το δεύτερο γύρο ερωτήσεων θα ήθελα ακόμα μία φορά να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε το χρόνο και αν είναι δυνατόν να υποβάλλετε όχι παραπάνω από δύο ερωτήσεις στη συνάδελφο, γιατί και ο χρόνος των απαντήσεων θα ξέρετε πολύ καλά ότι εξαρτάται και από τον αριθμό των ερωτήσεων. Ο κύριος Γκάρνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ καλά και σημαντικά αυτά που είπατε για το Πακιστάν. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα follow-up μετά τις ε, εκλογές. και με υπογραφή συμφωνίας να ενισχύσουμε περαιτέρω τη δημοκρατική δομή. Όσον αφορά το Αφγανιστάν, αναρωτιέμαι αν ο συνάδελφος ε, Μοριών ε, μπόρεσε να ε, εφαρμόσει τις ε, τεχνικές παρατήρησεις ε, στις εκλογές ώστε να διασφαλιστεί ε, η ποιότητα. Δεν έχω αποκτήσει οριστική εικόνα για το θέμα αυτό. Τι έχετε εσείς να πείτε. Και επίσης όσον αφορά την, τις γειτονικές μας χώρες. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε με την Ουκρανία διαπραγματεύσεις. Σύντομα θα, υπάρξουν, σύντομα θα πραγματοποιηθούν εκλογές. Προβλέπετε φέτος να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή. Πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Τηρήσατε τους χρόνους. Ρότσεκ. Αλλά θέλω να σας πω τώρα έχει κλείσει ο κατάλογος των παρεμβάσεων. 16-1. Εάν άλλοι θέλουν να παρέμβουν θα το κάνουν κάποια άλλη χρονική στιγμή. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία για το Ιράν. Είπατε ότι οι Αμερικανοί και εμείς θέλουμε να προωθήσουμε το διάλογο, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ε, με τον εμπλουτισμό ουρανίου και τις εκτοξεύσεις ε, πυράβλων. Θα ήθελα να μιλήσω για την κοινωνία των πολιτών στο Ιράν, διότι φοβάμαι ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μιλάμε μόνο για κυρώσεις και ξεχνάμε αυτή την πτυχή της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα το σχολιασμό σας. Και η δεύτερη ερώτηση έχει ως εξής. Υπάρχουν πολύ θετικές εξελίξεις ως προς τη σχέση Τουρκίας με την Αρμενία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να κάνουμε ίσως κάτι περισσότερο. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρότσεκ. Κέλαμ. Ευχαριστώ. Σημερίζομαι τις ανησυχίες σας ως προς τα ανησυχητικά νέα για το Ιράν. Και τα τελευ τις τελευταίες ημέρες ο παγκόσμιος τύπος ε, αμαυρώνει πολύ περισσότερο την εικόνα. Υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις. Εσείς μας είπατε ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο των κυρώσεων, αλλά φαίνεται ότι μέχρι τώρα το καθεστώς του Ιράν ε, θεωρεί ότι προτρέχει και εμείς απλώς τους ακολουθούμε και αντιδρούμε. Ίσως ε, σε μερικά χρόνια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση. Το σκεφτήκατε αυτό ότι το Ιράν θα έχει όπλα μαζικής καταστροφής καθώς και πυράβλους Πώς θα αντιδράσουμε τότε. Η δεύτερη επιλογή είναι πιο θετική. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό 20 χρόνια πριν κανένας δεν ήταν έτοιμος ε, να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση θα αποσυνδεθεί και θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Βλέπουμε λοιπόν ότι και το καθεστώς στο Ιράν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Θα επανέλθω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Ρότσεκ. Τι θα κάνουμε με την κοινωνία των εθνών στο Ιράν. Πώς μπορούμε να τους δώσουμε πολιτική και ηθική υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφος Μπότσκουρτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας με την Λατινική Αμερική. Αναφερθήκαμε στην κατάσταση στην Ονδούρα. Μιλάμε για μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική μέχρι τούδε. Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που προβλέπετε. Βλέπουμε εικόνες στην τηλεόραση σε τι αλγινή κατάσταση βρίσκεται ο λαός, ο ντόπιο ε, πληθυσμό. Μιλήσαμε για τους ε, πρεσβευτέ, για τους πρέσβει, για πώς ε, αντέδρασαν. Μετά είπαμε ότι ίσως θα υπήρχε ένα διαφορετικό είδος εκπροσώπησης αλλά δεν έγινε καμία αμνία για αυτή την, σε αυτή την τεχνική συμφωνία για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο Αρίας στις διαπραγματεύσεις του. Μπορείτε να είσαστε πιο σαφείς στην περίπτωση της Ονδούρας. Ευχαριστούμε. Μπροκ. Δύο λεπτά. Ε, ε, Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου δύο σύντομες ερωτήσεις. Καταρχήν, Αφγανιστάν. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Τα προβλήματα με τις εκλογές δείχνουν ίσως τα όρια που υπάρχουν στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Αρχικός στόχος ήταν να πάμε στο Αφγανιστάν για να βγάλουμε εκτός λειτουργίας την Αλκαΐδα. Μήπως θα άξιζε τον κόπο να ξανασκεφτούμε την κατάσταση να ξανακοιτάξουμε τους στόχους και να δώσουμε τέλος ε, στο θέμα. Δεύτερον, στο θέμα των πυράβλων και του αφοπλισμού, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις ε, και όσον αφορά την Τσεχία, το Ιράν, την Πολωνία, αλλά και όσον αφορά γενικά το θέμα του αφοπλισμού. Ε, δεν είναι πια τόσο μεγάλη η πίεση όσον αφορά τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ποιες είναι οι συνέπειες για την πολιτική γειτονία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι περιθώριο έχουμε για να κερδίσουμε κατανόηση της ρωσικής πλευράς. Ευχαριστώ. La parola Ευχαριστώ. δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ μία ερώτηση προς την Επίτροπο για το Ιράν. Ε, το Ιράν μας ξεγελάει εδώ και χρόνια. Έχουμε νέες ε, αποδείξεις ότι έχουν ε, πυρηνικά όπλα. Τι κυρώσεις θα μπορούσαμε να τους επιβάλλουμε ε, για να τους ασκήσουν πιέσεις. Γιατί υπάρχουν, υπάρχει μια πλειάδα κυρώσεων. Επίσης, ε, θέλουμε οι Παλαιστίνοι να ζουν μια φυσιολογική ζωή, αλλά το να καταπολεμηθεί και, ο, και η τρομοκρατία στην περιοχή και αυτό είναι βασικός στόχος. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γι' αυτό. Και ο Σελάγια στις Ονδούρες είναι ο πρώτος ο οποίος ε, ε, έθεσε τέλος στη συνταγματική τάξη. Αυτό δεν ήταν ο λόγος για να γίνει πραξικόπημα. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το να γίνουν οι εκλογές στο τέλος του χρόνου, τον Νοέμβριο. Κιλ Νίλσεν. Ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει ακόμα τεθεί για την Επιτροπή Έρευνας στο ΟΗΕ υπό την αιγίδα του Richard Κόλστον. Ε, που έδωσε την έκθεσή της για τα γεγονότα του Ιανουαρίου 2009 ε, στη Γάζα. Ε, εκεί υπάρχουν πράξεις που μοιάζουν με εγκλήματα πολέμου και σε ορισμένε περιπτώσεις με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχει ε, διαπράξει αυτά τα εγκλήματα. Και ζητούμε από το Ισραήλ να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα ε, με βάση τα διεθνή κριτήρια για αυτές τις παραβιάσεις και μέσα στους επόμενους έξι μήνες να δοθούν τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και επίσης να, δου, να δούμε πώς θα διώξει τους υπεύθυνους στο εβραϊκό κράτος ε, για τα εγκλήματα πολέμου. Επίσης έγιναν πάρα πολλές παραβιάσεις από το Ισραήλ και αναφέρονται στην έκθεση ε, θα πρέπει να σταματήσει η πολιορκία της Γάζας και να απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι και κυρίως τα πολυάριθμα φυλακισμένα παιδιά καθώς και τα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου. Ξέρουμε τι έγινε σε ανθρωπιστικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν τα βάσανα του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Το θέμα όμως, το ερώτημα που θέλω να σας θέσω κυρία Επίτροπε είναι τι κάνατε εσείς, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των σχέσεών της με τις Ισραηλινές αρχές ούτως ώστε να συμμορφωθούν με τις προσδοκίες ε, της Επιτροπής αυτής έρευνας του ΟΗΕ. Τι θα κάνει το Συμβούλιο. Θα ασχοληθεί, θα λάβει αυτή την έκθεση, το ελπίζουμε, ούτως ώστε να ξεκινήσει η αρχή του τέλους της εποχής της ατιμορρησίας, όπως την ονομάζω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και κλείνει ο δεύτερος γύρος των παρεμβάσεων με τον συνάδελφο Βανόρντεν ο οποίος θα μιλήσει για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την Επίτροπο. Χαίρομαι που ακούω θετικές παρατηρήσεις για τις διατλαντικές σχέσεις. Θα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό σε ερώτηση για τη Σρι Λάνκα, η οποία ζει μια πολύ δύσκολη περίοδο προσαρμογής μετά την ε, ήττα των τρομοκρατών ITTT. Βεβαίως ε, θέλουμε να υπάρχει γενεοδορία από την κυβέρνηση προς τους Ταμίλ και τους Ταμίλ που ζούσαν σε περιοχές ε, που προηγουμένως έλεγχε το ITT. Φυσικά υπάρχουν ανησυχίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις ε, ανησυχίες στα στρατόπεδα, όπου δέχονται ανθρώπους από τις πληγήσεις περιοχές. Ε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε το λαό της ε, Σρι μέσω της ε, δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησής του. Αλλά αντί να το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι του δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο τη ζωή. Νομίζω ότι παίζουμε και εμείς το σκοπό του LTT και τα όσα λέει η διασπορά η οποία επηρεάζεται από όσα λένε οι LTT Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δίνουμε περισσότερη βοήθεια, πιο πολύ ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσουμε ε, το δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στη Ριγλάνκα και στις δυτικές δημοκρατίες. Πώς μπορούμε να είμαστε πιο παραγωγικοί και πιο θετικοί απέναντι στη Ριγλάνκα. Ευχαριστώ τον κύριο Βανόρτεν. Και τώρα η Επίτροπος για το δεύτερο γύρο. Ε, ε, για να απαντήσω στον κύριο Γκάλερ. Νομίζω ότι ο στρατηγός ε, Μοριγιών προσπάθησε να εφαρμόσει την ίδια μέθοδο. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα προς Νότο και Ανατολάς. Αυτό το ξέρουμε εξ αρχής. Και καταφύγαμε, μάλλον προσφύγαμε σε, στους Αυγανούς πάνω από 8.000 που είχαν στρατευτεί, αλλά εν πάση περιπτώσει στο Νότο η ε, συμμετοχή του εκλογικού σώματος ήταν πολύ περιορισμένη σε σχέση με το Βορρά. Διαπιστώσαμε πράγματι ότι υπήρξαν πολλές παρατυπίες και το μόνο δυνατό και εφικτό θα ήταν οι Αυγανοί να θέσουν σε εφαρμογή και να εφαρμόσουν τους κανόνες που ενέκριναν οι ίδια. Αυτό ακριβώς απέτησε και ο στρατηγός Μοριγιών. Δηλαδή η Επιτροπή αυτή ε, που ασχολήθηκε με αυτές τις προσφυγές να τις εξετάσει. Η εξέταση δεν έχει λήξει και όταν θα γίνει κάτι τέτοιο θα μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα περιθώρια και να δούμε κατά πόσο ο πρόεδρος Καρζάη εξελέγει ήδη από τον πρώτο γύρο ή θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή ότι χρειάζεται ένας δεύτερος γύρος. Επίσης, να δούμε κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με την κυβέρνηση. Πολλές ιδέες υπάρχουν επιτάπητος, δεν είναι παρά ιδέες. Ίσως θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι θα είχαμε τον πρόεδρο, ως πρόεδρο, πρόεδρο τον ίν πρόεδρο Καρζάη και Πρωθυπουργό τον Αμπτουλάχ Αμπτουλάχ. Εν πάση περιπτώσει ήμουνα σε στενή επαφή με τον κύριο Μόρι ο οποίος επέδειξε μεγάλο θάρρος και εκείνος και η ομάδα του έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο αυτή. Ως προς την Ουκρανία, εδώ και δύο ημέρες στη Νέα Υόρκη έγινε η συνάντηση της Τρόικα, δηλαδή ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ουκρανία. Και είδαμε πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις, πώς έχουν εξέλιχθει. Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών θα μπορέσει να, να ισχύσει, να προωθηθεί. Ελπίζουμε όμω μέχρι το τέλο τη χρονιάς να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πολιτικό κομμάτι. Θα υπάρξει συνάντηση κορυφή ε, πριν τα Χριστούγεννα και αυτό ε, θα ασκήσει πίεση και στι δύο πλευρέ. Ε, και έχετε δίκιο, μετά έχουμε πάλι εκλογέ. Το αν μπορούν πριν τις εκλογές να πραγματοποιηθούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μάλλον δεν είναι πολύ πιθανό και νομίζω ότι και οι Ουκρανοί το βλέπουν αυτό ρεαλιστικά όσον αφορά το θέμα της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν. Να σας πω κύριε Ρότσεκ ότι πράγματι όσο μπορούμε προσπαθούμε να διατηρούμε διάλογο, να συνεχίζουμε το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών του Ιράν. Επικεντρωνόμαστε σε όχι ευαίσθητα θέματα όπως τα ναρκωτικά και τους πρόσφυγες όπου υπάρχει ε, κοινό ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, και από τη δικιά μας ε, και από την πλευρά του Ιράν. Υπάρχουν ε, και άλλα προγράμματα ε, σκοπεύουμε να ε, προοδεύσουμε σε θέματα όπως είναι η τηλεόραση και ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, το κανάλι στα Φαρσί και την ανταλλαγή φοιτητών. Το πρόγραμμα Erasmus Mundus είναι ανοιχτό και στους Ιρανούς και από καιρό σε καιρό να έχουμε επισκέψεις δημοσιογράφων και να συνεργαζόμαστε και μη κυβερνητικούς φορείς. Αυτό το κάνουμε στο βαθμό που μπορούμε. Θα θυμάστε ότι ο κύριος Μιγκαρέλη, ο αναπληρωτής ε, γενικός διευθυντής μου, πήγε στο Ιράν για να για να προσπαθήσει να ανοίξει τα προγράμματα αυτά, να τα κάνει πιο ανοιχτά, αλλά αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την Ιρανινή πλευρά. Αυτό είναι ε, δύσκολο θέμα. Ως προς ε, την ε, Τουρκία χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι, ότι θα υπάρξει άνοιγμα ως προς την Αρμενία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διπλωματικές ανταλλαγές, αλλά όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει κατόπιν να επικυρωθούν προβλέπω ότι ό,τι γίνεται στο χαρτί δεν ε, θα ε, πραγματοποιηθεί αμέσως, αλλά είναι πολύ θετικό το βήμα αυτό και φυσικά θα πούμε στους ε, Αρμένιους και συναντήθηκα και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, θα θέλαμε να δούμε περαιτέρω βήματα ε, όσον αφορά το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπακ ανάμεσα στην ε, Αρμενία και το Αζερπαϊτζάν. Ε, ο διάβολος όμως βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες. Ως προς το Ιράν πάλι, κύριε Κίλαμ. Πράγματι το Ιράν μέχρι τώρα αποφάσιζε την ταχύτητα. Από την άλλη όμως είχαμε εκλογές. Πριν τις εκλογές όλοι ξέραμε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τώρα ξέρουμε πόσο δύσκολε ήταν οι εκλογέ και το όλο πλαίσιο τους, οι συνέπειε των εκλογών. Τώρα όμως θα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο. Όλοι θα χαρούμε να δούμε θετικά αποτελέσματα, παρότι ξέρουμε ότι θα αργήσουν. Για πρώτη φορά οι Ιρανοί απαντούν Φυσικά είναι μια πολύ γενική απάντηση, αλλά και για πρώτη φορά οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να κάτσουν να συνομιλήσουν με τους Ιρανούς. Αυτό μετά από 8 χρόνια είναι αλλαγή στάσης και αυτό πάντα το ζητούσαν οι, Ιρανοί. Είναι θετικό βήμα. Ας δούμε τι θα τι θα κερδίσουμε με τους ε, διαλόγους αυτούς. Ε, υπομονή, δεν θα έχουμε υπομονή ατελείωτη, αλλά ετοιμάζουμε κυρώσεις, για παράδειγμα πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση θεωρήσεων. Αυτές οι κυρώσεις θα προετοιμαστούν, εξετάζουμε το θέμα, αλλά Ας αρχίσουμε να εφαρμόζουμε μια νέα πολιτική που έχει συζητηθεί, δεν έχει παρουσιάσει καρπούς μέχρι τώρα όμως. Και έχετε δίκιο ότι είδαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στην ε, κοινωνία του Ιράν. Εσείς ε, μπορεί να γνωρίζετε καλύτερα από μένα πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ε, υπό μεγάλη πίεση. Βλέπετε πώς η καταπίεση υπάρχει και για μένα είναι πολύ δύσκολο να πω εάν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μπορούμε να οδηγηθούμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Είμαστε δημοκράτες όμως. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει δημοκρατία. Ως προς την Ονδούρα. Κύριε Μπόσκουρτ. Τι κάνουμε συγκεκριμένα. Η συμφωνία σύνδεσης με την Ονδούρα δεν αποτελεί μέσο πίεσης. Όλες οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής και ιδιαίτερα η Κωνσταντίνα αλλά και άλλες θέλουν να πετύχουν τη συμφωνία αυτή και νομίζω ότι και οι Ισπανοί συνάδελφοι ελπίζουν επί προεδρίας τους ε, να έχουν, καλά αποτελέσματα. Πρώτα όμως θα πρέπει να λυθεί το θέμα με τις μπανάνες. Είναι δύσκολο εμπορικό το θέμα. Ε, χθες και προχθές είχαμε συναντήσεις με τις χώρες ΑΚΕ Τώρα θα πραγματοποιηθούν ε, διαπραγματεύσεις με τις ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και ο, Πανα... και ο Παναμάς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο ε, κ. Άστον επίσης πήγε στην Ουάσιγκτον διότι εμπλέκεται και η Τσικίτα στο θέμα. Είναι εμπορικό το θέμα, δεν είμαι επίτροπο εμπορίου, αλλά είναι εμπορικό το θέμα και κατόπιν θα επανέλθουμε στο πολιτικό θέμα. Υπάρχουν ε, διάφορες λύσεις που θα μπορούσε να εξετάσει κανεί. Η μία λύση θα ήταν να μην συμμετέχει η Ονδούρα. Άλλη λύση θα ήταν μια ρεαλιστική λύση που θα συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρέ, Αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος. Ε, μάλιστα ε, έγινε η ειδική συνάντηση για το θέμα αυτό. κύριε Μπρόκ, όσον αφορά το Αφγανιστάν, η ιδέα να διχάσουμε τους Ταλιμπάν ακολουθεί αυτήν την παλιά κατεύθυνση. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τους ε, ακραίους Ταλιμπάν. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Ταυτόχρονα δεν θα ήταν δυνατόν και δεν θα ήταν και σωστό να ε, αποσυρθούμε από το Αφγανιστάν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μετά ε, τις εκλογές ακόμα περισσότερο καθότι δεν γνωρίζουμε ε, κατά 100% το αποτέλεσμα. Στην ενισχυμένη αυτή στρατηγική θα πρέπει να προχωρήσουμε με πιο συντονισμένο τρόπο, ώστε να σταθεροποιήσουμε τη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επικεντρωθούμε περισσότερο από την νωρίτερα, όχι στην ε, στρατιωτική πλευρά, αλλά στην ε, πολιτική πλευρά. Άλλοι εταίροι δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα αυτό, αλλά τώρα αναγνωρίζουν το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούν με την πλευρά αυτή. Επίσης, δεν ε, είδαμε ακόμα πολύ θετικές ε, συνέπειες ε, στην πολιτική γειτονία από τον αφοπλισμό. Τώρα μόλις ξεκίνησε αυτό το θέμα του αφοπλισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Αυτό όμως οικοδομεί εμπιστοσύνη και ελπίζουμε αυτή η εμπιστοσύνη που έχει δημιουργηθεί και από τη δική μας πλευρά να έχει θετικές συνέπειες ε, ρωτήσατε επίσης, ε, κύριε Βανάλεν, ε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι, τι κυρώσεις προβλέπουμε. Ναι, μίλησα για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων ναι, και για τις θεωρήσεις. Θα το σκεφτούμε περαιτέρω. Ως προς τη Μέση Ανατολή, οι Παλαιστίνη, ε, υπό τον πρόεδρο Αμπάς έχουν δείξει ότι προσπάθησαν να πετύχουν καλά αποτελέσματα. Φυσικά πάντα μπορεί να κάνει κανείς περισσότερα, αλλά αυτό από την Ισραηλινή πλευρά οδηγεί σε, ε, σε πάυση της ε, επίκησης και αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε να πετύχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, όπως είπε και ο κύριος Πέτερινγκ. Ως προς τον Ζελάγια και το θέμα των, της Ονδούρας. Ναι, πρέπει να γίνουν εκλογές και έχετε δίκιο, οι εκλογές μπορεί να αποτελέσουν λύση, αλλά το θέμα είναι υπό ποιε συνθήκε. Ε, και η διεθνή κοινότητα ε, το σκέφτεται ακόμα, το ε, εξετάζει. Η συμφωνία... Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα αποτελέσει λύση, να υπάρχει διάλογος δηλαδή, αλλά όπως γνωρίζετε μια ή μια πλευρά, μια ή άλλη αρνείται το διάλογο. Δυστυχώ δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Σίγουρα δεν θα είμαστε παρατηρητέ στι εκλογέ αυτέ, αυτό είναι σαφέ. Όσον αφορά την έκθεση Goldstone. Αυτή η έκθεση θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Γενέβη. Σήμερα μάλιστα, 29 Σεπτεμβρίου. Δεν άκουσα τίποτα ακόμα για αυτό το θέμα και έχουν πολύ σημασία τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη λογοδοσία και θα καταπολεμήσουν την ατιμορρησία των, του ανθρωπιστικού, σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρωπιστικού δικαίου κτλ. Το τελευταίο ερώτημα αφορούσε τη Στριλάνκα του κυρίου Φανόρντεν. Καταρχάς, δουλέψαμε μαζί με την ε, Στριγλάνκα, συνεργαστήκαμε, δεν σταματήσαμε την ανθρωπιστική βοήθεια, εξακολουθούμε να βελτιώσουμε τις, ε, τις συνθήκες των εσωτερικά ε, με, μετατοπιστέντων ανθρώπων, των εσωτερικά εκτοπισμένων. Ε, παράλληλα όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο βλέπουμε ότι συχνά παραβιάζονται και αυτό είναι σαφές. Και επομένως πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα. Θα πρέπει εμείς να δείξουμε μια πιο επικοδομητική στάση, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα γεγονότα. Έχω προσπάθει να κάνω ό,τι μπορώ για τη Σρι Λάγκα. Αλλά συχνά δεν εισακούστηκα στην Επιτροπή των Συμπροέδρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο. Θα θέλαμε τώρα να συμπιέσουμε ακόμα περισσότερο το χρόνο, αντί για δύο λεπτά, ενάμιση λεπτό, για να σεβαστούμε το χρόνο που έχει στη διάθεσή της ε, η Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω πρώτος ομιλητής ο κ. Κούκαν. Μία ερώτηση. Μιλήσατε για τη σημασία τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατινική Αμερική και πώ θα αναπτυχθεί και θα καλλιεργηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Λατινική Αμερική δεν είναι μία ομοιογενή περιφέρεια. Υπάρχουν διαφορετικέ κυβερνήσει, χώρε κτλ. Παραδείγματο χάρη Βενεζουέλα. Ο, ο, ο Η νέα μελλοντική στρατηγική για την ε, συνεργασία με την ε, λατινική σχέση έλαβε υπόψη αυτό. Ξέρω ότι δεν μπορεί να υπησέλθετε σε βαθιές αναλύσεις τώρα, αλλά οποιοδήποτε σχόλιο είναι πρόσδεκτο. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Σεβαστήκατε και το 1,5 λεπτό. Ο κύριος Ομπιόλς, επίσης 1,5 λεπτό. Ο απολογισμός των σχέσεων ε, με την Λατινική Αμερική είναι θετικός και λαμβάνουμε υπόψη το δικό σας ε, ρόλο βεβαίως που ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Ε, αν ανακεφαλαιώσουμε τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι θεαματικές οι εξελίξεις. Έχουμε με το Μεξικό και τη Χιλή δύο συμφωνίες σύνδεσης και υπάρχουν και τρεις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με υποπεριφέρειες που λειτουργούν ε, πολύ αργά, με αργούς ρυθμούς. Και οι προβλέψεις είναι ανησυχητικές. Η μέθοδος περνώντας από μία ε, ολιστική στρατηγική σε υποπεριφέρειες, κάτι το οποίο είναι, είναι κάτι το θαυμαστό, περάσαμε σε ε, ορισμένα άκαμπτα σχήματα και νομίζω ότι ζούμε μία διαπραγμάτευση ε, όπου ακολουθείται αντίστροφη ε, στα αντίστροφη πορεία. Δεν νομίζετε ότι έφτασε η στιγμή να προβούμε σε μία ρύθμιση αυτής, αυτού του απολογισμού. Αρλάκη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ την κυρία Μπενίτα Φερέρο Μπάλτνερ που είναι παρούσα. Θα ήθελα να μιλήσω καταρχήν για τον αφοπλισμό. Όταν μιλάτε, όταν μιλήσετε για το θέμα του αφοπλισμού, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών πρόσφατα μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία το θέμα του Αφγανιστάν ε, βεβαίως μας είπατε ότι θα είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε ότι υπάρχει ευρέως ε, διαδεμένη διαφθορά σε αυτή την κυβέρνηση και ο αδελφός του Προέδρου, ο πρώην Υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης και ένας πρώην στρατηγός ε, είναι γνωστοί σε, στη διεθνή κοινότητα ότι προωθούν τα ναρκωτικά. Και λαμβάνεται αυτό, λαμβάνεται αυτό υπόψη όταν έχουμε δικούς μας στρατιώτες που διακινήραν τη ζωή τους. Τάνοκ, για ένα μισή λεπτό, ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, Επίτροπο και θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα προσέγγισης ε, Τουρκίας-Αρμενιστάν. Εγώ προήλθα από την ε, πρεσβεία του Αρμενιστάν και ο πρέσβης θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο της ε, Τουρκίας θα μπλοκάρει αυτή την προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε αυτή την, τη διεθνή συνθήκη διότι θα καταφέρουμε να ξεμπλοκάρουμε μια κατάσταση αστάθειας στο Νότιο Κάφκασο. Στο παρελθόν μου είπατε ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει ως προς την εφαρμογή ενός ε, προγράμματος στον Αγκόρνο Καραμπάχ για να προωθήσουμε την κοινωνία των ε, ε, πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται καθόλου εκεί. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς για τον Αγκόρνο Καραμπάχ έτσι ώστε να σταθεροποιήσουμε τον Νότιο Κάφκασο. Χτες ήρθα από την Κρυμαία και ως προς την Ουκρανία θα ήθελα να πω δεν υπάρχει ε, δυστυχώς καμία παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί ε, υπάρχει ε, σοβαρή παρουσία των Ρώσων και νομίζω ότι και οι Κινέζοι θα καλύψουν τα χάσματα εκεί. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς ε, να προβάλλουμε την παρουσία μας στην Κρυμαία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα ως προς την ΕΖΕΣ. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας για τις ε, μεγαλύτερες χώρες της ε, Ασίας, στην Νότια Ασία. Losing, 1,5 λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, Entschuldigung. Λάθο κουμπί πάτησα, συγγνώμη. Κυρία Επίτροπε, απαντήσατε ήδη σε πολλέ ερωτήσει ε, για την Ονδούρα. Ωστόσο, δεν έχω καταλάβει την βασική σας θέση για το πραξικόπημα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας ρωτήσω, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο πραξικόπημα ποια είναι. Ε, θα το ε, καταδικάσουμε και αν ναι θα υπάρξει ψήφισμα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν όχι γιατί όχι. Αναφέρθηκαν κυρώσεις, οι οποίες όμως είναι πολύ θόλες και αόριστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να... Ε, να ε, απελάσει τους ε, διπλωμάτες από την Ονδούρα. Και ε, η υποστήριξη προς τις αρχές που στήριξαν το πραξικόπημα θα θα παγώσει και αν όχι γιατί όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βάιγκολ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα σλοβένικα είναι δύσκολη γλώσσα, αλλά είναι επίσημη γλώσσα, άρα μπορώ να τα μιλήσω. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έρθει, έρθουν οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Εθνών και θα συντηθούν με τους βουλευτές. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τις εθνικές μειονότητες. Για την ε, σλοβένικη μειονότητα στην Καρίνσα που θα έρθει σε επαφή με σλοβένους εκπροσώπους και αυστριακούς. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε η Αυστρία να δεχθεί τις αρχές της δικής της νομοθεσίας που σέβεται, που αναγνωρίζει μάλλον την ε, σλοβένικη μειονότητα και ότι έχει κάποια δικαιώματα. Ευχαριστώ. Μενέντες βάλε για 1,5 λεπτό. Κυρία Φεραίρο Βάλτνερ, καταρχήν θα ήθελα και πάλι να σας συγχαρώ στην αρχή αυτής της θητείας, διότι δείχνετε καλή θέληση, βρίσκεστε εδώ και το κάνετε με μεγάλη πεποίθηση ως προς το θέμα του Ιράν. αν διαραγούν οι σχέσεις και οι διαπραγματεύσεις, έχετε πληροφορίες για το τι κυρώσεις θα μπορούσαμε να ε, επιβάλλουμε. Δεν θα επιμείνω στο θέμα της Κίνας και της Ρωσίας και το ρόλο τους, το σχολιάσατε. Γιατί ε, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της Ινδίας ως προς τις κυρώσεις. Ως προς τη διεθνή πειρατεία, ιδιαίτερα στον Ινδικό ωκεανό, ε, θα ήθελα να ρωτήσω, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες ε, κυρώσεις των κρατών μελών, τι πληροφορίες έχετε ως προς την σοβαρότητα του προβλήματος και την ε, δυσμενή ενδεχόμενα εξέλιξη του στο μέλλον. Ωραία. Κλείνει η συζήτηση. Την τελική απάντηση θα μας την δώσει η Επίτροπος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μια πληθώρα κρατών στη Λατινική Αμερική. Δεν πρόκειται για ένα ομοιογενές σχήμα, πρόκειται για διαφορετικές κυβερνήσεις. Αυτό που κάναμε ήταν το εξής. Προσπαθήσαμε να ε, έχουμε μία κατά περίπτωση προσέγγιση ανάλογα με την κάθε χώρα μέσα στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής και αυτό συμπληρώνει και την περιφερειακή προσέγγιση με την διμερή διάσταση. Δηλαδή ακριβώς αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Ε, κύριο Μπιόλς, έχετε δίκιο. Πολλές φορές οι διμερείς συμφωνίες ήταν πιο επιτυχής από τις περιφερειακές. Από την άλλη πλευρά όμως, οι περιφερειακές ε, συμφωνίες για πρώτη φορά ε, ασχολήθηκαν με τις περιφέρειες στην ολότητά τους, όπως ε, παραδείγματος χάρη για τις χώρες της ε, Λατινικής Αμερικής και τις χώρες των Άνδεων. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στον Δούρα, στην Ικαράγουα, είχαμε δει και τη Βολιβία ε, μέχρι τώρα όμως είχαμε υπερβεί τις δυσκολίες. Ακόμα και αν δεν ισχύσει κάτι τέτοιο υπάρχει μία ευελιξία ιδιαίτερα ως προς τις χώρες των Άνδεων είδαμε ότι μετά το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων αποφασίστηκε να έχουμε ε, μία ε, διτή προσέγγιση με βάση την ενημέρωση του πολιτικού διαλόγου Λακάν το 2003 και της διαπραγμάτευσης ε, μιας πολυμερής, ε, και στα πλαίσια μιας πολυμερούς ε, διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να βρισκόμαστε και μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Έτσι θεωρούμε ότι ότι ο τελικός στόχος είναι μία πλήρης πολυμερή σχέση μετά από έξι γύρους. Ο τελευταίος έγινε στις 21, 21 25 του μηνός με την Κολομβία και το Περού. Η Βολιβία δεν συμμετείχε και μια άλλη χώρα αποσύρθηκε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι μια επιτυχής σύναψη συμφωνήσαμε για το καθεστώς για την μπανάνα στη Γενέβη και ξέρουμε ότι η Κολομβία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το επιτύχουμε. Αυτό σημαίνει ότι αν πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, το κάνουμε. Και το ίδιο ισχύει και με την Ονδούρα αν δούμε ότι μετά αφού διευθετηθεί το θέμα του εμπορίου της μπανάνας η ονδούρα αποτελεί πρόβλημα, θα βρούμε μια ευέλικτη λύση, θα αλλάξουμε την εντολή και θα τα συμπεριλάβουμε τα υπόλοιπα. Αλλά χαιρόμαστε ότι, γιατί ως προς τον Ισημερινό, ο Ισημερινός επανέρχεται στις διαπραγματεύσεις και αυτό είναι πολύ θετικό. Δύσκολο βέβαια, αλλά προσπαθούμε να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Ως προς το Αφγανιστάν, γνωρίζω, κύριε Αλάκη, ο... και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι το θέμα της κυβέρνησης είναι ζωτική σημασίας και ότι η διαφθορά δυστυχώς αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη μάστιγα Γι' αυτό ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για το σύστημα δικαιοσύνης για να έχουμε μία νέα τάξη πραγμάτων ε, ως προς το δικαστικό σώμα τους εισαγγελείς και τους δικαστές, αλλά θα πρέπει να αποφαστεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτοί που πραγματικά είναι διεφθαρμένοι, να μην παραμένουν καθεστώς ατιμορρησίες. Ως προς το μέτωπο Τουρκίας-Αρμενίας, Ελπίζω, όπως είπε και ο κύριος ε, Τάνοκ, να υπάρξει επικύρωση, αλλά θα πρέπει να τους ε, ενθαρρύνουμε με ένα ψήφισμα. Ως προς το θέμα της κοινωνίας των πολιτών, στον Γκόρνο Καραμπάχ, θα ήθελα να πω ότι εγώ προσπάθησα να βοηθήσω αυτά τα προγράμματα, αλλά υπάρχουν προσκόμματα εδώ και εκεί μεταξύ των συμβαλωμένων μερών ο κύριος Σέμνεπη και μία ομάδα αξιωματούχων μετέβη εκεί. Από τη μία πλευρά ήταν δύσκολο, μάλλον και από τις δύο πλευρές το ζήτημα ήταν δύσκολο. Το ανέφερα και στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είχαμε καλή έκβαση. Όταν ήμουν στο Αζερμπαϊτζάν θυμάμαι ότι μίλησα με τον ίδιο τον πρόεδρο για να δώσω όλες τις δυνατότητες. Αλλά δυστυχώς πάντα υπάρχουν συμφέροντα στη μέση των με ή τον δε. Να μην υπάρχει πλήρης ε, ε, σύμπνοια ή συμφωνία. Κάτι είπε ο κύριος Τάνοκ ε, εκτός μικροφώνου. Ίσως έχουν άλλο καθεστώς φορολόγηση. Σε πάση περιπτώσει καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ως προς την Ουκρανία είχα μία αντιπροσωπεία από την Κρυμαία τέσσερις-πέντε εβδομάδες πριν και συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Γιούσενκο να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την Κρυμαία αλλά χρειάζεται χρόνος. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά που προείπατε. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες, περισσότερο παρόντες στην Κρυμαία για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολη. Ως προς την Ινδία, ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, είναι πάντα πολύ δύσκολη μια τέτοια ε, συμφωνία. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου είναι πιο δύσκολες γιατί υπάρχει μια κατάσταση δούνε και λαβίν πολύ δύσκολη. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την Ινδία ως στρατηγικό εταίρο. Θα γίνει διάσκεψη κορυφής με την Ινδία και όλα αυτά τα ζητήματα θα και θα πρέπει πριν από τη διάσκεψη να δούμε πόσο έδαφος έχουμε καλύψει. Η Ινδία διαδραματίζει όλο ένα και μεγαλύτερο σημαντικό ρόλο, αλλά είναι επιφυλακτική ως προς το θέμα έφνης των κλιματικών αλλαγών, όπου δεν είναι παρούσα, όπως θα θέλαμε στην Κοπενχάγη. Τέλος, κυρία Λέζιν, ως προς το θέμα της Ονδούρας, η θέση μας είναι πολύ σαφής. Έχουμε ε, καταδικάσει εδώ και καιρό την, ε, ε, το πραξικόπημα, έχουμε παγώσει τις ε, πολιτικές επαφές, όλες τις επαφές με τους διπλωμάτες, την κυβέρνηση de facto δηλαδή έχουμε, τις έχουμε παγώσει και έχουμε αναστείλει όλα τα προγράμματα με την κυβέρνηση. Δεν έχουμε παγώσει αυτά που αφορούν την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε κάνει λοιπόν ακριβώς αυτά και στον κύριο Βάγκλ να πω ότι ως προς τις ε, εθνικές ε, μειονότητες ε, ξέρετε ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται και από τις δύο πλευρές όμως. Και Αν μάλιστα Δελβάγε, όσον αφορά το Ιράν, νομίζω ότι είπα ότι θα, μπορούσε να, θα μπορούσαν οι ε, να είναι πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων, η απαγόρευση θεωρήσεων. Ε, υπάρχουν και άλλες ιδέες, ε, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα όμως. Και ω προς την πειρατεία, να πω ότι είναι ένα νέο τρομακτικό φαινόμενο. Ποιο θα το σκεφτόταν αυτό πριν λίγα χρόνια. Σημαντικό όμως είναι να καταπολεμούμε όχι μόνο την πειρατεία ε, την υπεράκτια πειρατεία, αλλά ε, και στις ακτές μας ε, και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε και ο Λουί Μισελ και η Κάρελ Τεχούστ το κάνουν αυτό στις σομαλικές ακτές. Έχουμε τεράστια προγράμματα, όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με την εκρίζωση της στόχιας, κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Χαίρομαι όμως που βλέπω ότι ήδη πολλοί Ευρωπαίοι εργάζονται στην Αταλάντα που είναι μία πρώτη ευρωπαϊκή δράση συνεργασίας ε, στη θάλασσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Ήταν πολύ ευρία η συζήτηση, άγγιξε διάφορα θέματα. Μπήκατε σε πολλές λεπτομέρειες παρά τον περιορισμένο χρόνο και θεωρώ ότι ικανοποίησατε τους περισσότερους συναδέλφους. Αλλά προκαλέσατε σίγουρα και τον ενδιαφέρον κυρίως για θέματα τα οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ελπίζω ότι αυτή η συνεργασία που είδαμε την έκφανσή της σήμερα μεταξύ ημών να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, Σταματάμε τώρα και θα ξαναρχίσουμε στις 5 ε, η ώρα μια κοινή συνεδρίαση με την αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτική Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Μολδαβία. Με μια ανταλλαγή απόψεων με τον Πρωθυπουργό τη Μολδαβία, τον Βλαντ Φίλατ. 15 λεπτά διάλειμμα. Συνάδελφοι, θα ήθελα να καθίσετε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε με ακρίβεια. Είναι εδώ ο Πρωθυπουργό ο Βλάντ Φίλατ. Ήρθε στην ώρα του με ακρίβεια. Συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας. Σήμερα Έχουμε ως μαδικό σημείο στην ημερήσια διάταξη το πολύ σημαντικό θέμα της ακρόασης των δύο αυτών Μολδαβών κυρίων. Η συνάδελφος, η Μόνικα Μακβέη, είναι η πρόεδρος της αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Ελπίζω αυτή η συνεργασία που ξεκινά σήμερα να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, είναι μεγάλη τιμή για μένα και για τους συναδέλφους να σας υποδεχτώ εδώ, να υποδεχτώ αυτή την πολύ σημαντική αντιπροσωπεία. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ανανεώθηκε πρόσφατα ε, και υπάρχουν πολλές προσδοκίες γιατί μόλις μία εβδομάδα πριν ε, δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνη σε εσά και υπάρχει μεγάλη προσδοκία λοιπόν γύρω από την κυβέρνησή σας. Είναι η πρώτη κυβέρνηση της ε, Μονταβίας που βγήκε από την τροχιά της ε, ΕΣΔ. και είναι η πρώτη μη κομμουνιστική κυβέρνηση μετά την κομμουνιστική περίοδο. Αυτό είναι μια ψηφίδα της ε, ιστορίας της Μολδαβίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζουμε την θέλησή σας για ανανέωση, την θέλησή σας να μπείτε και να συμμετάσχετε στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Μεταξύ των σημείων που θα ήθελα να αναφέρω, σημείων του προγράμματός σας, ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για τη χώρα σας και για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν ο στόχος να διαλυθεί το κρατικό μονοπόλιο ή τα κρατικά μονοπόλια. Και μετά την οργανωμένη οικονομία της κομμουνιστικής εποχής ε, έχετε τη θέληση να εγκαθιδρύσετε μια οικονομία της αγοράς, να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, διεθνών ε, επενδυτών, παραγόντων, τόσο ώστε να προσελκυστούν κεφάλαια στη χώρα σας, να ανανεώσετε την αγροτική οικονομία, να βελτιώσετε τις σχέσεις συνεργασίας με τις όμορες χώρες, κυρίως με τη Ρουμανία, και να επιλύσετε τα εναπομείναντα εδαφικά προβλήματα. Εμείς ε, χαιρόμαστε για αυτή τη θέληση ανανέωσης και κύριε Πρωθυπουργέ θα θέλαμε να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε ούτως ώστε αυτές οι προκλήσεις να υλοποιηθούν και η χώρα σας να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, σε αυτή τη νέα πατρίδα που είναι η Ευρώπη. Αυτά και σας δίνω χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση το λόγο κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω ρουμανικά. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας πέρασε ένα χρονικό διάστημα αρκετά δραματικό. Διένυσε μία δραματική φάση και πορεία. Όπως είπατε, πρόκειται για την πρώτη κυβέρνηση της Κισινάου που είναι μη κομμουνιστική. Και αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ και που μπόρεσα να προβώ τη, στη σύσταση κυβέρνησης. Όπως ξέρετε, ο κύριος Λέγκου και εκείνος συμμετείχε στην πρώτη κυβέρνηση της Κισινάου που προέβη σε ένα πλήρως πρόγραμμα και δημιουργήσαμε μία, ελπίζουμε, σταθερή κυβέρνηση. Δυστυχώς, μετά από τις μεταρρυθμίσεις εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων και δυστυχώς έφτασε επικεφαλής με μεγάλη πλειοψηφία. Όπως ξέρετε, οκτώ χρόνια, για οκτώ χρόνια, μας κυβερνούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο πρόεδρος ήταν ο Βορόνιν, ο οποίος ε, προέβη στη σύσταση μιας κυβέρνησης δορυφόρου της ε, Ρωσίας. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν μια πολύ δυσχερή κατάσταση στη δημοκρατία μας, διότι έπρεπε να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες, οι βασικές, οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Ξέρω ότι πολλοί από εσά παραστήκατε και παρευρεθήκατε στο Κισινάου. Είχαμε πολλά μέλη τα οποία παρευρέθηκαν με βάση τη συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Μολδαβίας. Είχαμε μονοπόλιο της οικονομίας. Ο τύπος δεν είχε βασικές ελευθερίες, δεν υπήρχε ελευθεροτυπία και ένα εκατομμύριο πολίτες έπρεπε να φύγουν από τη χώρα. Και αυτό έγινε και για πολιτικούς λόγους και για να μπορέσουν να βρουν θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν άνοιξαν τα σύνορά μας. Παρόλο ότι συμμεριζόμαστε τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Θα πρέπει να αναφέρω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο χαρακτήρισε την κομμουνιστική κυβέρνηση. Και αναφέρομαι στη ρουμανοφοβία. Υπήρχε εχθρική στάση έναντι της ε, ε, Ρουμανίας, ιδιαίτερα σε σχέση με το καθεστώς των θεωρήσεων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Όμως, το πιο δραματικό χρονικό διάστημα είναι το διάστημα μετά τις εκλογές της 5ης Απριλίου, όταν άρχισαν οι διαμαρτυρίες στο Κισινάου, όταν υπήρξε ένα συγκεκριμένο κίνημα με θύματα, με ανθρώπινα θύματα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι βασανίστηκαν, κλείστηκαν στη φυλακή και δεν αναγνωρίστηκε η κυβέρνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, αποτέλεσε υποστήριξη για την κοινωνία του Κισινάου και έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα να αντισταθούμε. Βεβαίως, θα πρέπει και χρειάστηκε να γίνουν πρόορες εκλογές και θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό είχε οικονομικές συνέπειες. Είχαμε λοιπόν πρόορες εκλογές στις 29 Ιουλίου και είχαμε και παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με λιγότερη ή περισσότερη νοθεία, περισσότερες ελευθερίες θα θέλαμε να πιστεύουμε, από όπου ανέκυψε μια δημοκρατική κυβέρνηση που απαρτίζεται από τέσσερα κόμματα, μη κομμουνιστικά κόμματα, τέσσερα κόμματα κοινοβουλευτικά που αποτελούν την Συμμαχία για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Την προηγούμενη Παρασκευή εξελέγει και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και συστάθηκε κυβέρνηση την προηγούμενη Παρασκευή. Βεβαίως θα πρέπει να διανύσουμε μεγάλο χρονικό διάστημα για να λειτουργήσουν αυτοί οι θεσμοί και αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για τον, την εκλογή του Προέδρου της ε, Μορδαβίας. Για να εκλεγεί Πρόεδρος χρειάζονται 61 έδρες. Εμείς έχουμε 53, άρα χρειαζόμαστε 8 ψήφους επιπροσθέτως. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλες εντάσεις και ε, ελοχεύει εκ νέου κίνδυνος πρόωρων εκλογών. Οι πρόωρες εκλογές δεν μπορούν να λάβουν χώρα για δεύτερη φορά. Και άρα θα πρέπει να διενεργηθούν εκλογές του χρόνου, γιατί δεν μπορούν να διενεργηθούν πρόορες εκλογές δύο φορές μέσα στο ίδιο έτος. Αυτή είναι η κληρονομιά που μας άφησαν οι κομμουνιστές, που διακυβέρνησαν τη χώρα. Έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα άνευ προηγουμένου. Στο τέλος του έτους θα φτάσει το 20,5% του ΑΕΠ. με συγχωρείτε, το 12,5%. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία δυσμενή περίοδο κατά τη διάρκεια αυτής της εκλογικής διαδικασίας και από την άλλη πλευρά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ υψηλές δαπάνες, ένα υψηλό κόστος που πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες με βάση την θριαμβολογία που είχαν προωθήσει οι κομμουνιστές στο Κισινάου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από πού προέρχεται αυτό το έλλειμμα, ποια είναι η πηγή αυτών των χρεών, των οφειλών που πρέπει να καταβληθούν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αναγνώριση λύσεων και πόρων για να χρηματοδοτήσουμε αυτό το δημοσιονομικό έλλειμμα για να μπορέσουμε να καταβάλουμε μισθούς ε, καθώς και συντάξεις. Και αναφέρομαι εδώ στην διακυβέρνηση επί 8 έτη από τους κομμουνιστές οι οποίοι δεν θα πρέπει να μπορούν να θριαμβολογούν και να λένε ότι διακυβέρνησαν δημοκρατικά. Εμείς βασιζόμαστε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπερβούμε τις δυσχέρειες αυτές. Και εδώ αναφέρομαι όχι μόνο στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και για τις γενικότερες προοπτικές που θα πρέπει να γνωρίσουν οι Μολδαβοί πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μου επιτρέπετε, ε, είχα προετοιμάσει ε, έναν λόγο, αλλά θεώρησα ότι δεν είναι σκόπιμο να σας τον εκφωνήσω. Θα ήταν σκοπιμότερο να απαντήσω σε ενδεχόμενες ε, δικές σας ερωτήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια, ένας ουσιώδης διάλογος και ευελιξία. Θα, σας, ε, θα απαντήσω με μεγάλη χαρά στις τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον στο συνάδελφο που είναι πρόεδρος της ε, Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας, Μόνικα Μακοβέη. Ευχαριστώ συνάδελφοι και κύριε Πρωθυπουργέ. Θα περάσω στα ρουμανικά. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποια σύντομα σχόλια πρώτα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι υπήρξε μεγάλη συμμαχία σε σχέση με τις εκλογές του Απριλίου, κάτι το οποίο είναι ύψης της σημασίας, θα πρέπει να παραμείνετε ενωμένοι έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στο κυβερνητικό σας πρόγραμμα και για να εφαρμόσετε τις μεταρρυθμίσεις έχετε τη δική μας υποστήριξη για την έγκριση και τη θέση σε εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η χώρα. Θα αναφερθώ σε μερικές από αυτές, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία και βεβαίως μέτρα για, την, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει ανεξάρτητη τηλεόραση και ραδιόφωνο, ανεξαρτησία των ΜΜΕ, κράτος δικαίου, κοινωνία των πολιτών, καθώς και άλλες πρακτικές όπου ε, παντού χρειάζεται ελευθερία κινήσεων. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει ένα θαύμα εν μία νυχτή. Νομίζω ότι ε, έχετε εξηγήσει στους πολίτες σας ότι πρέπει να είσαστε ρεαλιστές και και για τους δικούς σας πολίτες και για εμάς, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για τις μεταρρυθμίσεις και αυτό διαμέσου μέτρων που θα ληφθούν άμεσα για να προγραμματίσετε τις μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη συνάντηση όπου δεν θα μπούμε εν λεπτομερία σε θέματα, αλλά θα ήθελα να σας δώσω μία συμβουλή, να έχετε συγκεκριμένα σχέδια για κάθε τομέα όπου θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε και ο πληθυσμός και τα ευρωπαϊκά όργανα να μπορέσουν να σας παρακολουθήσουν πού θέλετε να φτάσετε, με τι μέσα, ποιο είναι το κόστος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να πληρωθούν αυτοί οι στόχοι χρειάζεται χρειάζεται σαφήνεια και προβλεψιμότητα σε αυτή την ε, μεταβατική περίοδο της χώρας. Είμαι πεπισμένη ότι έχετε κατά νου όλα αυτά τα μέτρα από κοινού με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, όπως ορίζουν τα σχέδια δράσης. Θα ήθελα να σας πω ότι έχετε τη δική μας υποστήριξη και το λέω για άλλη μια φορά. Έχετε τη δική μας υποστήριξη για μια νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένω στο γεγονός ότι η διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ύψη της σημασίας για τις αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν στην υποψήφια χώρα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε πολύ καλά με αυτή τη διαδικασία και τις αλλαγές. Και κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο, έμπρακτα, θα ήθελα το Κοινοβούλιο της ε, Δημοκρατίας της Μολδαβίας να ορίσει μια επιτροπή εξωτερικών έτσι ώστε να συσταθεί μια επιτροπή συνεργασίας με το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θαυμάσια η παρέμβασή σας. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Πάσκου. Ευχαριστώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας συγχαρώ διότι κερδίσατε τις εκλογές σε αυτή την κυβέρνηση συμμαχίας και με μεγάλη μας χαρά να συνεισφέρουμε και εμείς αυτή τη μεγάλη σας νίκη. Οι προσδοκίες της κυβέρνησης είναι πολύ υψηλές και προέρχονται και από τον πληθυσμό ο οποίος ζει και διάγει δύσκολο βίο. Βεβαίως ε, ξέρουμε τι έγινε με τις πρώτες εκλογές, με την πρώτη αναμέτρηση και αποστολή μας είναι να μπορέσετε εσείς να ανταποκριθείτε στην οικονομική κατάσταση και τις ε, οικονομικές δυσχέρειες. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στους συναδέλφους σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, ότι η βασική μεταρρύθμιση είναι να λύσετε τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός, όπως είπε και η πρόεδρος της αντιπροσωπείας, δηλαδή να υπάρξει ένας προγραμματισμός και η πρώτη σας φροντίδα είναι να αντιμετωπίσετε τη δυσμενή κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Στη συνέχεια θα πρέπει να ευεργητηθείτε και από ένα διάλογο με τους ε, κομμουνιστές, διότι μόνο με μια κυβέρνηση συνεργασίας θα επιληθεί η λύση, η οποία πλήττει όλους τους ε, Μολδαβούς. Σε σχέση με τη διεθνή συγκυρία, πέρα από τις εσωτερικές εντάσεις που αντιμετωπίζετε, θα πρέπει να βασιστείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι Μολδαβοί περιμένουν τη δική μας υποστήριξη και θα την έχουν και εκφράζουμε την ελπίδα ότι εάν δεν υπάρχει καλή θέληση από τη Ρωσία, τουλάχιστον να είναι η δέτερη, ουδέτερη η Ρωσία, έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στο δύσκολο καθήκον σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πάσκου. Ο κύριος Βέμπερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό για τα νέα του καθήκοντα και για την εξέλιξη στη δυσμενή κατάσταση της Μολδαβίας. Θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ συμμετείχα στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διενέργεια των εκλογών και ήθελα να σας πω ότι με εξέπληξε η υπεποίθηση των ανθρώπων ότι η ψήφος τους μετράει και μπορεί να ορίσει μια πραγματική αλλαγή. Και πιστεύω ότι οι Μολδαβοί αξίζουν αυτή την αλλαγή. Βεβαίως αντιμετωπίζεται μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και δεν θα ήταν ε, ευχάριστο για μια τέτοια δύσκολη κατάσταση να βρεθείτε σε μία νέα προεκλογική εκστρατεία αν ξαναγίνουν πρόορες εκλογές. Αν φτάσετε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κερδίσετε ξεχωριστά αυτές τις εκλογές διότι γνωρίζουμε πώς διενεργούνται οι εκλογές συνήθως. Αλλιώς η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική με βάση το, τα ΜΜΕ, διότι πολύ λίγοι γνώριζαν ότι εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα υπήρχε και κάτι άλλο αν παρακολουθούσαμε τα ΜΜΕ, όπως βλέπαμε από τη διεθνή τηλεόραση. Εάν φτάσετε σε αυτή την κατάσταση που ελπίζω να αποφευχθεί, ο δικός μας ρόλος σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν να πείσουμε τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα ότι δεν υπάρχει αστάθεια στη δημοκρατία της Μολδαβίας, αλλά πρόκειται για ένα διαδικαστικό θέμα το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί διαφορετικά. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, πέρα από το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της ε, Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ένα πρώτο βήμα προς εσάς θα ήταν να αλλάξουμε το καθεστώς των θεωρήσεων για τους πολίτες της Μολδαβίας. Και η Επιτροπή ΑΘΕΤ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών καθώς και η αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλλον και Δημοκρατίας της Μολδαβίας θα μπορέσει να ζητήσει την αλλαγή αυτού του καθεστώτος έτσι ώστε οι Μολδαβοί πολίτες να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρόκειται για μια μαζική έξοδο των Μολδαβών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που ήθελαν μέχρι τώρα ήδη βρίσκονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα πρέπει να γνωρίζει αυτό το κοινοβούλιο ότι κανείς ε, βρίσκεται στον τόπο του, το σπίτι, ο χώρος διαμονής είναι κάτι το διαφορετικό για τον καθένα από εμά και ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα κύματα μετανάστευσης για εξέβρεση εργασίας και γι' αυτό ακριβώς θα σας βοηθήσουμε. Θα πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα. Οι Μολδαβοί που θα ε, μπορούν να μεταβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα επιστρέφουν στην πατρίδα τους, θα μπορέσουν να μεταφέρουν τις ευρωπαϊκές αξίες στην πατρίδα τους και έτσι θα αλλάξει και η νοοτροπία που ίσχυε στη, στη Μολδαβία μέχρι τούδε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λέζιν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις έχω σχετικά με την ουδετερότητα της Μολδαβίας. Στο άρθρο 11 του Συντάγματος ε, αναφέρεται ε, ακριβώς αυτή η ουδετερότητα. Σύμφωνα με ε, εκθέσεις που ακούσαμε, βελτιώνονται οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ καθώς και στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης για την ειρήνη. Θέλετε να γίνετε μέλος ε, του ΝΑΤΟ. Και μία ε, προσχώρηση σε, ε, σε μια οργάνωση όπως είναι το ΝΑΤΟ δεν αντίκειται ακριβώς στη ρήτρα αυτή της ουδετερότητας. Επίσης, αναφέρατε ότι θέλετε όσο πιο σύντομα προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στρατιωτική ένωση. Η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε κάποιο κράτος μέλος, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν ε, να βοηθήσουν ε, να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ε, για να το βοηθήσουν. Αυτό ε, στο άρθρο 42.7 τη συνθήκη της Λισαβόνα. Αυτές ήταν οι ερωτήσει. μου. Ευχαριστώ. Είναι γεγονό ότι η κατάσταση στη Μολδαβία προβλέπει ουδετερότητα αλλά βεβαίως και το Σύνταγμα προβλέπει ότι θα πρέπει να αλλάξει το, το δίκαιο αυτό, δηλαδή το δικαιοδοτικό πλαίσιο για τους πολίτες. Θέλουμε ε, να προβάλλουμε εμβαθυμένες σχέσεις με το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να διανύσουμε ένα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες τι σημαίνει ΝΑΤΟ. Γιατί βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών θεωρεί ότι πρόκειται για μια εχθρική συμμαχία γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρωσικός ε, τύπος δέσποζε στη χώρα μας. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κακή θεώρηση της Ατλαντικής ε, Συμμαχίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ότι υπάρχει μία ε, σταθερή σχέση μέσα στα πλαίσια της περιφέρειάς μας και θα πρέπει οι πολίτες να αποφασίσουν ποιο θα είναι το στάτους δημοκρατίας της Μολδαβίας και επ' αυτού του θέματος. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί καταφέρατε να εκλέξετε μία κυβέρνηση υπέρ της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι καταφέρατε να ακυρώσετε τη θέληση του προηγούμενου καθεστώτος που είχε προβάλει το καθεστώς των θεωρήσεων και το οποίο είχε επιβάλει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα είναι η μελλοντική σχέση Ρουμανίας και Δημοκρατίας της ε, Μολδαβίας και πώς θα εγγυηθείτε την ελευθεροτυπία, διότι στο παρελθόν ο τύπος βρισκόταν στα χέρια πολύ λίγων και, και δεν υπήρχε ελεύθερος τύπος. Σεβερίν. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένες υποδείξεις και ερωτήματα. Το πρώτο μήνυμα προέρχεται από αυτή την ε, αίθουσα. Σήμερα μιλάμε πολύ ρουμανόφωνοι, αλλά το θέμα της Μολδαβίας είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι στο μέλλον θα διατρανώσουμε αυτή τη θέληση ότι δηλαδή χρειαζόμαστε τη δημοκρατία της Μολδαβίας όχι σαν γειτονικό κράτος αλλά σαν ευρωπαϊκό κράτος. Και αυτή η σχέση θα πρέπει να αποτελέσει μέλημα όλων και όχι μόνο μερικών μελών του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, η συμμαχία σας είναι η συμμαχία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης, για την ενσωμάτωση στην Ευρώπη και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Πιστεύετε ότι η προευρωπαϊκή σας δέσμευση θα πρέπει να ε, ορίζεται μέσα στα πλαίσια μιας θέλησης υπέρ της Μολδαβίας, δηλαδή να δημιουργήσετε μια οικονομική και κοινωνική καθώς και περιφερειακή συνοχή, καθώς και πολιτισμική, έτσι ώστε να έχετε έναν κοινό δημόσιο χώρο, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να αποφαίνονται ελεύθερα και να φτάσετε σε μια κοινή ελάχιστη ατζέντα. Το τρίτο μήνυμα αφορά την αντιπολίτευση δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Μολδαβίας. Θα πρέπει να τους πούμε ότι συμμετέχουν στο πλουραλιστικό σύστημα της μολδαβικής κυβέρνησης, όπως ισχύει σε κάθε δημοκρατία, αλλά υπάρχει το δέλεαρ να προβάλλουν ένα αντάρτικο κατά της ε, κυβέρνησης κάτι το οποίο θα τους απομακρύνει από τον πολιτικό χώρο. Άρα σας ενθαρρύνουμε να δημιουργήσετε μία πολιτική συνοχή με διάλογο και με την αντιπολίτευση, να ενθαρρύνουμε την αντιπολίτευση, να ταχθεί υπέρ του διαλόγου και να μην υπονομεύσει την κυβέρνηση του Κισινάου. Και η τελευταία ιδέα έχει ως εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση κατεπηγόντως θα πρέπει να ε, εγκρίνει ένα, θέμα, ένα συγγνώμη, πρόγραμμα οικονομικής αρρωγής προς την ε, δημοκρατία της ε, Μολδαβίας. Μπορούμε να σας δώσουμε οποιαδήποτε συμβουλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά αν δεν έχετε μαζική οικονομική αρρωγή από εμάς, μαζί με την κοινοπολιτεία της Ρωσίας ή με άλλα κράτη, τότε δυστυχώς θα διατρέξετε μεγάλο κίνδυνο γιατί η φτώχεια δεν βοηθάει τη δημοκρατία. Ονορεύολε Μπουζόη. Μπουζόη. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα πολύ θετικά αποτελέσματα, διότι από τη Δευτέρα έχουμε να κάνουμε μια πραγματική δημοκρατική κυβέρνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει την προσέγγιση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος. Θα έπρεπε να καταδείξετε ένωση τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, προσπάθησε να υπονομεύσει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου με μία ψήφο και Δείξατε μεγάλο θάρρος. Καταφέρατε λοιπόν να κερδίσετε όχι μόνο εσείς αλλά και οι πολίτες της ε, Μολδαβίας. Βρισκόσαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο κατάφερε να αλλάξει η στάση μας έναντι της δημοκρατίας της ε, Μολδαβίας, διότι υπήρξε μεγάλη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Επιτροπή δεν ήταν ε, ένθερμος οπαδός σας ή υπέρμαχος των ε, θέσεων σας. Ξέρουμε ότι υπήρξε νοθεία, υπήρχε βία, υπήρξαν βασανιστήρια και βεβαίως η οικονομική κατάσταση είναι το πιο δυσχερές ε, ζήτημα. Χρειαζόσαστε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς αναμένουμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την ε, δράση σας. Θα ήθελα να σας απευθύνω τρεις ερωτήσεις. Τι θα αλλάξει ως προς την πολιτική σας προσέγγιση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, κάτι που ανησυχεί τους ευρωπαϊκούς εταίρους. Θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο μπορείτε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των σύνορων και τι θα γίνει με την υπερνηστερία. Ξέρουμε πώς έχετε κινηθεί μέχρι τώρα, αλλά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κατά πόσο θα δεχτείτε μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση της ειρήνης στην υπερδνηστερία. Λίζερ. Ε, e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρωθυπουργό, δεν είμαι, Πρωθυπουργέ, δεν είμαι ε, Ρουμάνος. Θέλω να επιβεβαιώσω όμως ότι έχετε την υποστήριξη όλων μας, όλων όσων είμαστε σε αυτή την αίθουσα και όλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πριν από λίγους μήνες ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Πολωνία και έκανα ένα λάθος. Δέχτηκα ε, στην πατρίδα μου εκπροσώπου σας, μίλησα με τους ε, Πολωνούς μου και είπαμε ότι ίσως θα πρέπει να περιμένουμε επαορίστο ε, για να έρθουν κάποιες εκλογές. Αλλά έκανα λάθος εκτίμηση. Ευτυχώς. Θα ήθελα να σας θέσω κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Η ιστορία μας μοιάζει με τη δική σας. Αυτό που σας περιμένει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με βάση τις αναλύσεις ε, η δημοκρατία της ε, Μολδαβίας, αν δεν λάβει εξωτερική βοήθεια, δεν θα μπορέσει να εξέλθει από την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και οι Ηνωμένε Πολιτείε δήλωσαν ότι θα δώσουν μια κάποια οικονομική βοήθεια. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως πάνω απ' όλα είναι οι δηλώσεις που έγιναν ε, για τις πιστώσεις από τη Ρωσία. Η προηγούμενη κυβέρνηση μίλησε για αυτές. Αλλά είπαμε, υπόθηκε ότι υπήρχαν πολιτικές ε, προϋποθέσεις που συνόδευαν την ε, ε, χορήγηση των πιστώσεων. Ε, σε ό,τι αφορά την υπερνηστερία μάλιστα, θα ήθελα να, σας, να μου πείτε ποιες είναι οι απαιτήσει της κυβέρνησής σας και η στάση της κυβέρνησής σας απέναντι στη Ρωσία. Λοιπόν, μετά από αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων, θα δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό. Ceea ce ține de relațiile cu România. Σε σχέση με, την, ε, με τη σχέση μας με τη Ρουμανία, η ιστορία έχει καταδείξει ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις ε, γειτονίας. Αυτό δείχνει και το παρελθόν και αυτό διαγράφει και το μέλλον. Τώρα τι κάνει ο τύπος στη δημοκρατία της ε, Μολδαβίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο νόμος ήταν κακός, η εφαρμογή του δεν ήταν σωστή και γι' αυτό οδήγησε στην κατάσταση που γνωρίζετε. Ιδιαίτερα σε σχέση με το οπτικοακουστικό σύστημα, τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο δεν υπήρξαν ε, ελευθερίες. Θα αλλάξει το καθεστώς στο εγγύς μέλλον έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει δημόσια τηλεόραση η οποία να πληροφορεί τους πολίτες και να μην τους χειραγωγεί. Ως προς ερωτήσεις του κ. Μπουσόη, μας μιλήσατε για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα γεγονότα του Απριλίου. Εμείς είχαμε ζητήσει την υποστήριξή σας διότι σας είπαμε τι συνέβη πραγματικά. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που θα ήθελε η αλήθεια να αναγνωριστεί από όλους. Τι διεμήφθη στην χώρα μας και από τη διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό έχουμε αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση και την επόμενη εβδομάδα θα συσταθεί Επιτροπή Έρευνας για να ζητήσουμε την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου που θα μας βοηθήσουν με εμπειρογνώμονες για την περίοδο που θα χρειαστεί. Δεν έχει οριστεί ακόμα. Θα πρέπει να συνταχθεί μία έκθεση ευραίος φάσματος για να γνωρίζει η διεθνής κοινότητα τι συνέβη, αλλά και οι πολίτες μας. Και έτσι ώστε εκείνοι που προέβαλαν αυτό το ιδεχθέ σενάριο να μην το προβάλλουν και στο μέλλον, να μην δηλαδή επαναληφθεί αυτή η τραγωδία. Θα πρέπει να φτάσουμε σε συγκεκριμένες ε, δράσεις και όχι σε δηλώσεις και θα ήθελα να σας πω ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Κύριε Σεβερίν, Μιλάμε για μια συμμαχία για την συμμετοχή και την ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Η διαδικασία βεβαίως ένταξης σημαίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Εμείς μιλάμε για την ευρωπαϊκή προσχώρηση, αλλά καταρχήν θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί άρδιν η δημοκρατία της Μολδαβίας και αυτό όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για τους δικούς μας τους πολίτες. Ως προς την ασφάλεια των σύνορων χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επίτροπης και ξέρετε ότι θα ε, υπάρξει μια αποστολή προς τα σύνορα ιδιαίτερα τα σύνορα Μολδαβίας-Ουκρανίας για να υπάρξει πραγματική αποτελεσματικότητα. Επίσης, στρατεύματα για την διατήρηση της ειρήνης. Αυτό το είχαμε προβάλει και στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ασφάλεια των σύνορων. Ως προς το θέμα της οικονομικής ε, αρρωγής από την ε, Ρωσία ε, έγινε λόγος για ένα πολύ υψηλό ποσό, έγινε λόγος δηλαδή για 500 εκατομμύρια και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και του κομμουνιστικού κόσματος. Δυστυχώς και χτες μάθαμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών έφτασε σε αυτό το καθεστώς των πιστώσεων χωρίς να γίνουν προηγούμενες διαπραγματεύσεις για να έχουμε μία οικονομική υποστήριξη για τα 15 επόμενα χρόνια από την κοινοπολιτεία της Ρωσίας, χωρίς να ξέρουμε ποιο θα είναι το πολιτικό κόστος. Διαβιβάσαμε αυτό το μήνυμα και μας ενδιαφέρει αυτή, αυτό το μεγάλο κονδύλι, αυτή η μεγάλη πίστοση. Έχουμε διαβάσει αυτά τα στοιχεία προς τη κοινοπολιτεία της ε, ε, Ρωσίας και όπως ξέρετε θα γίνει μια συνάντηση μέσα στον μήνα Οκτώβριο με τον, πρόεδρο, με, τον Πρωθυπουργό μάλλον συγγνώμη, με τον πρόεδρο Μετβέντεφ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε με επαγγελματισμό να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα σχέση χωρίς συναισθηματισμούς και θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι σχέσεις ε, θα τις διαχειριστούμε με αξιοπρέπεια. Θα τον Πρωθυπουργό για τις απαντήσεις του. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για τον διορισμό σας και για την ψήφο εμπιστοσύνη στο Εθνικό σας Κοινοβούλιο. Ελπίζω αυτή η προοπτική ένταξης να συγκεκριμενοποιηθεί πιο γρήγορα από ότι ίσχυσε για τη Ρουμανία, γιατί για μας η διαδικασία ένταξης κράτησε 10 χρόνια και κάτι. Τι μέτρα θα λάβετε για το δημοσιονομικό σας έρημα το οποίο είναι υπέρογκο και τι πολιτικά μηνύματα λαμβάνετε από τη Μόσχα μέσα στα πλαίσια αυτού του υπέρογκου δανείου που θα λάβετε. Και από όσο ξέρω, ε, να σας ρωτήσω τι θα γίνει με το μεταναστευτικό κύμα προς το εξωτερικό που υπάρχει από πλευράς Μολδαβίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας και τους συνεργάτες σας που δώσατε αυτή την ηρωική μάχη και οι Ρουμάνοι και οι Ολλανδοί φιλελεύθεροι στάθηκαν στο πλευρό σας στην προεκλογική εκστρατεία. η παράνομη κυβέρνηση της υπερνηστερίας παίρνει κάποιες οδηγίες από τη Ρωσία ή έχει κάποια αυτονομία. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνουμε για να βρεθεί μια λύση. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το θέμα της υπερνηστερίας. Ευχαριστώ τον κύριο Βαμπάλεν. Ο κύριος Σούλτς. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε ε, Υπουργέ Εξωτερικών. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας ε, να μεταρρυθμίσετε και να σταθεροποιήσετε την χώρα και να την φέρετε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ο ίδιος ότι υπολογίζεται να γίνουν πρόορες εκλογές την επόμενη χρονιά για να ε, λυθεί το θέμα αυτό της πολιτικής κατάστασης. Τι θα κάνετε για να ε, ενθαρρύνεται την ε, συμμετοχή στις εκλογές. Διότι από ό,τι κατάλαβα η συμμετοχή στις εκλογές ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σούλτς. Ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και καιρό είμαι υποστηριχτή ε, των ε, προσπαθειών της Μολδαβίας ε, να προσεγγίσουν την Ευρώπη και επικροτώ και τις προσπάθειες σας για δημοκρατία. Επέστρεψα χθες από την Ουκρανία, περιμένουν ένα πακέτο πολλών εκατομμυρίων από ε, την Κίνα που ε, αποτελεί θεόσταλτο δώρο για την ε, κυβέρνηση αλλά αποτελεί μεγάλο σοκ για τη Ρωσία. Από ό,τι κατάλαβα η Κίνα έχει υποσχεθεί και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και στην Μολδαβία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει και πώς βλέπει η Ρωσία τα μεγάλα αυτά χρηματικά ποσά που πηγαίνουν προς τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Κλείνει εδώ δεύτερος γύρος. Ξαναδίνω το λόγο στον Πρωθυπουργό πριν περάσουμε στον τρίτο και τελευταίο γύρο. Όπως ξέρετε, προβλέπεται και η σύναψη συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ξέρουμε ποιοι είναι οι δυσμενείς ε, όροι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παραμέτρους που είναι ιδιαίτερα αυστηρές, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο, γιατί αντιμετωπίζουμε μία δυσμενή πολιτική κατάσταση. Ξέρετε ότι συζητήσαμε το θέμα και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Ελπίσουμε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το πλαίσιο, γιατί διαφορετικά το κοινωνικό κόστος που θα πρέπει να καταβάλουμε θα είναι πολύ υψηλό και οι πολίτες δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν. Σας είπα ότι είναι μια διαδικασία διαπραγματεύσεων Στη συνέχεια θα συμφωνήσουμε, θα υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα δούμε στη συνέχεια τι θα διαμειφθεί για να χρηματοδοτήσουμε αυτό το δημοσιονομικό έλλειμμα. Πέρα λοιπόν από τις αρρωγές αυτές θα πρέπει να διορθώσουμε τον προϋπολογισμό, να περιορίσουμε τις δαπάνες και να αυξήσουμε τα έσοδα. Ποια είναι τα πολιτικά μηνύματα που λαμβάνουμε από την ε, κοινοπολιτεία της ε, Ρωσίας. Προς το παρόν δεν έχουμε μηνύματα. Παρακολουθούν την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Στις 7-8 Οκτωβρίου θα γίνουν δύο διαπραγματεύσεις στο Κισινάου. Θα μιλήσουμε με ευθύτατη γλώσσα και δεν θα θέλαμε να υπάρξει χειραγώγηση από πλευράς του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Κισινάου. Γιατί υπάρχουν μεμονωμένα συμφέροντα έναντι της ε, Μόσχας. Τώρα, τι θα γίνει με εκείνους που δουλεύουν στην Αλοδαπή θα πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα, αλλά υπό ποιου όρους θα πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μία συγκεκριμένη προοπτική. Θα πρέπει να μπορέσουν να διαβιώσουν και να εργάζονται στη χώρα τους. Τι θα γίνει με την υπερδνηστερία τώρα. Είναι αυτόνομη ή επηρεάζεται από το Κρεμλίνο όπως λέμε εμείς στην ιδιόγλωσσά μας. Δεν αποτελεί μυστικό για κανέναν ότι υπάρχει υποστήριξη από την κοινοπολιτεία της Ρωσίας, ιδιαίτερα ως προς το οικονομικό σκέλος, δηλαδή εκ νέου υπάρχει αυτή η χειραγώγηση και η χρηματοδότηση. Τι θα γίνει με τους πολίτες μας που δεν βρίσκονται στην χώρα. Θα πρέπει να βρούμε μία τελική λύση. Η καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρχει η ηλεκτρονική ψήφος, έτσι ώστε να υπάρχει και ασφάλεια και έλλειψη νοθείας. Θα πρέπει να ορίσουμε στην νομοθεσία μας ότι εκεί όπου εργάζονται Μολδαβοί πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέσω πρεσβείας ή προξενείου. Τώρα σε σχέση με την Κίνα. Και εμείς, ε, όπως ξέρετε, έχουμε συνάψει μια συμφωνία στα πλαίσια του κατασκευαστικού τομέα. Ζητήσαμε από τον νυν Υπουργό Οικονομίας να μας μιλήσει για αυτά τα κονδύλια που προβλέπονται. Θα πρέπει στη συνέχεια να διαλευκάνουμε το θέμα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν σωστές επενδύσεις στις υποδομές για να κατασκευαστούν έργα οδοποιίας, γέφυρες, κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν ε, προβλέπεται του παρόντος. Τώρα ως προς τις πιστώσεις ε, από την Κίνα ή την ε, Μόσκα θα προτιμούσαμε οι πιστώσεις αυτές να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να υπάρξει ένα άνοιγμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κισινάου. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τη συζήτηση. Είναι ο τελευταίος γύρος. Δεν μπορώ να δεχτώ άλλες παρεμβάσεις πέρα από τις πέντε που προβλέπονται. Κέλαμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να σας ε, στείλω θερμούς χαιρετισμού από την Εστονία. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι και ανακουφισμένοι ε, με τον σχηματισμό μιας ε, φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης στη Μολδαβία. Πολύ σωστά είπε η συνάδελφος ότι όλοι χρειαζόμαστε, όλοι θέλουμε η Μολδαβία να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον να είναι κομμάτι της Ευρώπης. Είχαμε πολλές χαμένες ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο λαός της Μολδαβίας ότι αξίζει στον λαό της Μολδαβίας καλύτερη ζωή και δημοκρατία. Είμαστε διτεθειμένοι να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε την ε, ανατολική εταιρική σχέση, ε, για παράδειγμα την διευκόλυνση για τις θεωρήσεις και επίσης ως προς την τρανσδνηστερία. Απαντήσατε, η ερώτησή μου όμως έχει να κάνει με την μακρόχρονη λαθρεμπορία όπλων. Μιλήσατε για τις προσπάθειες ελέγχου των συνόρων, να έχει σταματήσει το λαθρεμπόριο όπλων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάτσιν. Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι Ρουμάνος, δεν μιλώ Ρουμάνικα, ούτε Μολδαβικά. Θυμάμαι όμως την τελευταία θητεία που ήρθατε εδώ και Ρουμάνος σε συνάδελφος είπε ότι μιλάει πολύ άσχημα τη γλώσσα σας. Ε, σήμερα μιλάνε όλοι οι Ρουμάνοι ρουμάνικα σε εσά και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μεγάλο βήμα προόδου στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ε, Ρουμανίας και της Μολδαβίας. Θα ήθελα να ε, κύριε Φίλατε, να εκφράσω την εκτίμησή μου που ήρθατε τον Απρίλιο και ήρθατε και σήμερα και για να μας ε, μιλήσετε και να μας πείτε από πρώτο χέρι τις ε, εμπειρίες σας. Τολμηρό είναι αυτό που κάνατε. Καταφέρατε συνασπισμό των τεσσάρων μη κομμουνιστικών κομμάτων. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την νίκη σας και τη νέα θητεία σας. Ε, πρόκειται για δύσκολη θητεία. Πιο εύκολο είναι να κερδίσει κανείς τις εκλογές, ε, πολύ πιο δύσκολο είναι να κυβερνήσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να, γίνει πιο, να υπάρξει σταθεροποίηση στην ε, Μολδαβία. Κύριε, Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας καλέσω να είσαστε όσο γίνεται πιο ευέλικτος ώστε να ε, επιτευθεί η εκλογή Προέδρου. Ελπίζω να κυβερνήσετε σοφά, να στείλετε μήνυμα προς όλους τους ανθρώπους ε, στη Μολδαβία ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Κάποιες ερωτήσεις ε, σχετικά με την οικονομική κατάσταση στη χώρα σας. Νομίζω ότι το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι στη χώρα σας περιμένουν οικονομικά θαύματα εδώ και τώρα. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς οικονομικά θαύματα εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι όμως απόλυτα θεμητό η επιτυχία σας, η επιβίωσή σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεγγύη, μας. Θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν, ε, το Συμβούλιο, να βρουν τρόπους να υποστηρίξουν οικονομικά τη Μολδαβία, να προτείνουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο με μεγάλη χαρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, χωρίς ε, την βοήθεια αυτή δεν υπάρχει ελπίδα ούτε για μας ούτε για τη Μολδαβία. Κλείνοντας, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να πω ότι στην αίθουσα αυτή δεν υπάρχει κανείς που να μην υπερασπιστεί την ε, εδαφική ακαιρεότητα της Μολθαβίας συμπεριλαμβανομένης της Τρανσνιστερίας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, <clears throat> Κύριε Πρωθυπουργέ, πήγα μαζί με τους ε, συναδέλφους για να παρατηρήσω τις ε, εκλογές στο Κισινάου το καλοκαίρι στις αρχές του Μαΐου. Και μιλήσαμε και μεταξύ μαζί σας, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί θέλαμε να ακούσουμε την γνώμη σας. Ε, εκείνη την εποχή τίποτα δεν ε, προϊόνιζε ότι θα σας ξανασυναντούσαμε με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Φυσικά το ονειρευόμασταν, ε, φυσικά το συζητήσαμε, αλλά ήταν δικό σας όνειρο. Ε, κανένας εκείνη τη στιγμή δεν ήταν πεπισμένος ότι η συμμαχία σας θα οδηγούσε στην νίκη. Τώρα, το θέμα κλειδί, το ερώτημα κλειδί είναι οι προεδρικές εκλογές. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό. Και τώρα ένα επώδυνο ερώτημα. Επόδυνο για τη Μολδαβία, νομίζω τουλάχιστον. Είναι το δράμα που προέρχεται από το διχασμό της χώρας, το θέμα της υπερνηστερίας. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο παράγοντας που δεν επιτρέπει την επανένωση της χώρας. Ξέρουμε όλοι ποιο κρύβεται από πίσω. Ποιο είναι αυτό ο παράγοντα. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Σήμερα, μετά τις εκλογές, υπάρχει μια αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή στην κοινωνία, υπάρχει αλλαγή στον πληθυσμό σας. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο η εξουσία και η κυβέρνηση. Αυτό που έχει σημασία είναι και οι προσδοκίε του λαού, οι ελπίδε του. Και ένα άλλο ερώτημα η αντίδραση των Μολδαβών και κυρίως των νέων Μολδαβών που φύγαν στο εξωτερικό και που σήμερα γνωρίζουν τι τους προσφέρει μια δημοκρατία, τι μπορεί να τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που γνωρίζουν ότι υπάρχουν και άλλες ε, πρώην ανατολικές χώρες που στο μεταξύ εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι αυτό τους δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον. Φυσικά πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές αλλαγές πρώτα στη Μολδαβία. Αλλά νομίζω ότι η μη επαρκή συμμετοχή των νέων και των μεταναστών οφείλεται στο γεγονός ότι η μέρα των, των εκλογών έγινε μία αργάσιμη μέρα. Δεν μπόρεσαν να πάνε στην ε, Μολδαβία για να ψηφίσουν ήταν εργάσιμη μέρα η μέρα των εκλογών. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να το λάβετε υπόψη για τι επόμενε εκλογέ. για το μέλλον. Και μια άλλη ερώτηση. Εσεί, ω Πρωθυπουργό, πώ βλέπετε την ανατολική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα μέσα στα πλαίσια αυτή τη εταιρική σχέση που θεωρείτε εκ των όνου κάνευ. Ποια είναι τα μέσα τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Μολδαβία Φυσικά υπάρχει μια ολόκληρη πανοπλία από μέσα και εργαλεία που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν. Παραδείγματο χάρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε, αλλά και διάφορα κράτη θα μπορούσαν να σας βοηθήσουμε, μονομένα. Μια άλλη ερώτηση. Πώς βλέπετε τη σχέση σας με τη Ρωσία. Ποια είναι η γνώμη σας για την ε, καλή γειτονία με τη Ρωσία. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον ανατολικό γείτονα. Τι μπορείτε να κάνετε ούτω ώστε αυτός ο γείτονα να μην παρεμποδίσει τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Τι μπορείτε να κάνετε ούτω ώστε αυτός ο γείτονα να ενθαρρύνει τον εκδημοκρατισμό σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάη. Η κυρία Νικολάη. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις με κάθε σεβασμό και γνωρίζοντας ότι έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις. Είσαστε η πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση με πολλές προκλήσεις και σας εύχομαι κάθε τύχη. Πώς βλέπετε την κατάσταση της υπερδνηστερίας, πώς το βλέπετε σαν πολιτικό σχέδιο μακρόπνοα. Εσείς σας είπαμε τι επιθυμούμε, θα θέλαμε να ξέρουμε τι επιθυμείτε εσείς από μας. Πώς βλέπετε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο αναγκαία και πόσο γρήγορη πρέπει να είναι αυτή η αρρωγή διότι δεν γνωρίζουμε πολύ καλά την οικονομική κατάσταση της ε, Μολδαβίας και ποια είναι τα επίγοντα σχέδια όπου χρειαζόσαστε την υποστήριξή μας μέσα στα πλαίσια και της συνταγματικής μεταρρύθμισης διότι με το παρόν συνταγματικό καθεστώς βρίσκεστε εδώ και ένα χρόνο σε μία κατάσταση διαδοχικών εκλογών, κάτι το οποίο επιδεινούται σε αυτή την περίοδο κρίσης. Ευχαριστώ τον κύριο Νικολάη. Ουγγουρεάνου. Και εδώ κλείνει η συζήτηση με αυτή την τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, είχαμε ψηφοφορήσει σε μια άλλη επιτροπή στην οποία συμμετέχω. Μα εγκατέλειψε το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορία και καθυστερήσαμε. Εγώ σπούδασα στα αγγλικά και τώρα θα περάσω στα ρουμανικά. Θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ και εγώ για το γεγονός ότι άλλαξε και το καθεστώς θεωρήσεων έναντι των ε, Ρουμάνων πολιτών, κάτι το οποίο ήταν παράλογο. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω κατά πόσο ε, έχετε ένα πρόγραμμα για να ρυθμίσετε το γλωσσικό καθεστώς στη Μολδαβία. Ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα να σχολιάσετε είναι κατά πόσο μπορείτε να διευθετήσετε νόμιμα τα, πώς να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα γεγονότα του Απριλίου του 2009 ως προς τις ε, παρατυπίες που διαπιστώθηκαν από πολλούς παρατηρητές. Επειδή έχουμε και εκπροσώπους από την Κομισιόν εδώ, θα ήθελα να μας πείτε και να μας πούν πώς έχει η κατάσταση, πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μολδαβία, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την πραγματογνωμοσύνη μας και την αρρωγή μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση άμεσα, χωρίς διαμεσολαβητές. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Έκλεισε η συζήτηση και θα ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό με την τελική απάντηση. Σε σχέση με την ανατολική εταιρική σχέση, όπως ξέρετε, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της ε, Μολδαβίας και εκπρόσωπο πως της Δημοκρατίες της ε, Μολδαβίας συμμετείχε χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου. Τώρα έχουμε μία στεναρή θέση. Θέλουμε να εφαρμοστούν όλα τα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ανατολική εταιρική σχέση και θα ήθελα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της εμπορίας όπλων στην περιοχή της υπερνηστερίας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη επί του θέματος. Ως προς την υπερδνηστερία, πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να ρυθμιστεί το όλο ζήτημα με βάση το συνταγματικό Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιος θα είναι ο προπομπός της επίλυσης του ζητήματος και μιλώ για την αποστρατικοποίηση και την έλλειψη εγκλήματος στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορεί να λυθεί αυτή η διαφορά και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει μία διευθέτηση επεξηγώντας το ζήτημα στους Μορδαβούς πολίτες. Δηλαδή να υπάρχει μία σωστή επικοινωνία με ανθρώπους ε, της επιστήμης, του πολιτισμού, για να υπάρξει μία απότερη διευθέτηση και να, έχουμε, να μιλάμε για ένα ενιαίο, μία ενιαία γεωγραφική ενότητα πολιτών. Θα θέλαμε την άμεση υποστήριξή σας και για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας εγγυηθώ το ότι η δημοκρατία της Μολδαβίας θα προβεί σε δράσεις και δεν θα αρκεστεί σε λόγια ως προς τις ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιολογήσουμε αυτές τις προοπτικές έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στις δικές μας δεσμεύσεις και αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μήνυμα το οποίο να καταδεικνύει ότι οι Μολδαβοί πολίτες μπορούν να αναμένουν πολλά από τις προοπτικές αυτές συνεργασίες. Το πιο επίγον είναι η αρρωγή για τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Παράλληλα όμως θα πρέπει να γίνουν και επενδύσεις για έργα υποδομών, ιδιαίτερα ως προς τα διασυνοριακά προγράμματα. Έτσι ώστε να υπάρχει επικοινωνία πέρα από το γλωσσικό. Ξέρουμε τι καταστροφές έγιναν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταστράφηκαν πολλές γέφυρες πάνω από το Δούναβι και το Δνίστερο και οι πολίτες της Μολδαβίας για να πάνε στη Ρουμανία θα πρέπει να διατρέξουν 100 χιλιόμετρα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν κατασκευαστούν γέφυρες. Επίσης θα πρέπει να έχουμε πόσιμο νερό παντού στη Μολδαβία, κάτι το οποίο δεν ισχύει μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Και υπάρχουν ε, και θέματα υγείας και υγιεινής εδώ. Ε, μιλήσατε για το γλωσσικό καθεστώς. Το Σύνταγμα στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της ε, Μολδαβίας αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό καθεστώς. Αντιμετωπίσαμε μία ιδιάζουσα συγκυρία. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το γεγονός ε, ε, ότι οι Αμερικανοί μιλάνε αγγλικά σημαίνει και για μας ότι οι Μολδαβοί μιλάνε ρουμανικά μουτά της μουτάντης. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να επιληθεί σωστά και ειρηνικά. Ως προς τα γεγονότα της 5ης Απριλίου είπαμε ότι έχουμε αναλάβει δέσμευση έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε και να διαλευκάνουμε την κατάσταση όπως εξελίχθηκε με σημαντικές κυρώσεις, με αυστηρές κυρώσεις. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις και νομίζω ότι απάντησα σε όλες. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό. Εξαντλητικές ε, και πλήρες οι απαντήσεις. Αυτή η μεικτή συνάντηση με την αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Μολδαβία και την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ε, τελειώνει εδώ. Ε, θα κλείσουμε με τα σχόλια της συμπροέδρου της κυρίας Μακοβέη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει, θα ήθελα να διαβάσω στους συναδέλφους του Κοινοβουλίου ότι έχω καταγράψει όλα τα ζητήματα που ετέθησαν σήμερα θα τα εντάξουμε στην Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, επιθυμούμε έναν διαρκή και ανοιχτό διάλογο μαζί σας. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε σας βήμα, έτσι ώστε να μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και θα σας ενημερώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις εξελίξεις μας. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας γεωγραφικά είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Ε, μοιραζόμαστε τις ευρωπαϊκές αξίες και ελπίζουμε κάποτε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Θα τα πούμε αύριο στις 30 του μηνός στις 9 για την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων για το βραβείο Ζαχάροφ. Λύε τη συνεδρία.